Good morning everybody. Thank you for reminding me to... Καλή σας μέρα. Έχουμε αρκετά μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης στην αίθουσα. Καλώς ορίσατε. να την τη της συνεδρίασης. Έχετε στα χέρια σας το σχέδιο ημερησία διάταξης. Πριν, την... πριν υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάποιες αλλαγές που θα ήθελα να προτείνω. Ο κ. Βαλκάρθελ έχει σήμερα το πρωί δύο σημαντικές συνεδριάσεις ε, που σχετίζονται άμεσα με τις αρμοδιότητές του ως Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε δεν θα καταφέρει να έρθει εδώ πριν από το μεσημέρι. Ευτυχώς ο Γενικός Γραμματέας της CMR, ε, του Συμβουλίου των Δήμων και Περιφερειών ε, της Ευρώπης, που ήταν προγραμματισμένος για το απόγευμα, μπορεί να είναι εδώ και είναι μαζί μας σήμερα το πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πνεύμα συνεργασίας που δείχνει. Οπότε προτείνω δύο αλλαγές στο σχέδιο μέσα διάταξης η ανταλλαγή απόψεων με το Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης να λάβει χώρα σήμερα το πρωί αμέσως μετά την ε, ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Φιλ Βιν Owen από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και η συζήτηση της έκθεσης πρωτοβουλίας του κύριου Βαλκάθερ, Βαλκάθερ να περάσει για το απόγευμα μετά την παρουσίαση του ΕΣΠΟΝ από την πλευρά ΕΣΠΟΝ. Αν συμφωνείτε μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτή την αλλαγή. Ε, ο κ. Βανίστελ Ρόι, ε, τι ώρα θα ε, γίνουν οι ψηφοφορίες ε, πρόεδρος. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Οι ψηφοφορίες θα ξεκινήσουν λίγο μετά τις 11 και 4. Είναι λίγο περίπλοκο αυτό, περιπλέκει τα πράγματα για ε, τα μέλη. Ε, πρόεδρος, ε, ναι, χτες είχα ζητήσει να στάλει το χρονοδιάγραμμα, δυστυχώς δεν εστάλει, το αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα χτες. Ζητώ συγγνώμη, θα λυθεί το πρόβλημα, δεν θα ξανά... Θέλετε να λαμβάνετε γραπτό στο χρονοδιάγραμμα. Είμαι συντονιστής και έχω και άλλους συντονιστές, λέει, λέει ο κ. Βανίστελ Ρόι. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν και άλλες συνεδριάσεις και έρχονται να ψηφίσουν. Δεν μπορεί η γραμματεία να στείλει ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι, ασφαλώς. Παρακαλώ πολύ στείλτε το χρονοδιάγραμμα. So we can Ωραία, υιοθετούμε λοιπόν την ημερησία διάταξη. Τέλεια. Σημείο 2 της ημερησίας διάταξης. Έγκριση των πρακτικών. Το σχέδιο πρακτικών της συνεδρίασης της 15 Οκτωβρίου είναι διαθέσιμο ε, στο ίντερνετ. Στις 17 Σεπτεμβρίου αποφασίσαμε ως ε, μικρή συνεισφορά στην πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου ε, για μείωση της χρήσης του χαρτιού είχαμε αποφασίσει να μην διανέμονται τα πρακτικά. Αν δεν εκφραστούν αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις μέχρι το τέλος συνεδρίασης θα θεωρούνται τα πρακτικά ως εγκεκριμένα. Συνεχίζουμε με τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Έχω μία μόνο ανακοίνωση για σήμερα. Κύριε Μόρτζε. Euh, Θα ήθελα στα πρακτικά να αναφερθεί, να αναφερθούν οι παρατηρήσεις που είχα κάνει στο πλαίσιο της συνάντησης των συντονιστών σε ό,τι αφορά τον ειδικό ε, εισηγητή για την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Yes, you want Πρόεδρος, θα αναφερθεί στα πρακτικά η παρατήρησή σας. Στα πρακτικά μας δεν μπορούμε να αναφέρουμε την ε, παρατήρηση αυτή ε, στα, σε πρακτικά συνάντηση των συντονιστών. Θα αναφέρουμε αυτή σας την παρατήρηση όμως στο πλαίσιο των πρακτικών της ομάδας γιατί είχε γίνει και στην ομάδα σε παλιότερη συνεδρίαση. Περνάμε στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Έχω μία μόνο ανακοίνωση, όπως είπα και προηγουμένως. Το, η ομάδα υψηλού επίπεδου για την παρακολούθηση της απλοποίησης ε, των δικαιούχων ε, ε, του, της πρωτοβουλίας στρατηγικών επενδύσεων ε, στην πρώτη συνεδρίαση της ομάδας υψηλού επίπεδου για αυτής δηλαδή της ομάδας τα 12 μέλη της ομάδας και ο πρόεδρος κ. Κάλλας συναντήθηκαν με εκπροσώπους ε, των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Το Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύθηκε από την Επιτροπή Ρέτζι μέσω του κ. Ζέλαρ, Ζέλαρ τον Αντιπρόεδρο. Ο στόχος της ομάδας υψηλού είναι να μειωθεί η επίπτωση των ε, περίπλοκων γραφειοκρατικών κανόνων επί των δικαιούχων. Θα αντιμετωπίσει σημαντικά θέματα όπως ε, οι δυνατότητες μείωσης του κόστους, ε, πρόσβαση στα, στο Ταμείο πόρους ε, και το gold plating. η Επιτροπή μας υποστήριξε θερμά την σύσταση αυτής της ομάδας και πιστεύει ότι μέσω της απλοποίησης μπορούν να αρθούν εμπόδια και φραγμοί στην, και, να γίνουν αυτά τα κονδύλια διαθέσιμα σε ακόμα περισσότερες περιφέρειες και δικαιούχους. Ε, αναμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα της εργασίας ομάδας Ψιλοπέλ το συντομότερο δυνατό ε, μέσω μιας ανταλλαγής απόψεων με, τις, με την Επιτροπή Ρέτζι στο πρώτο εξάμεινο του 2016. Αυτή είναι η ανακοίνωση, η μοναδική μου ανακοίνωση και περνάμε στο πρώτο ε, ουσιαστικό σημείο της Μέσης Διάταξης σήμερα, ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Phil Wayne Owen, ε, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, σχετικά με την ειδική έκθεση ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου ε, 10 10-2015 με τίτλο «Φάλματα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής για την συνοχή». Οι δημόσιες συμβάσεις παίζουν ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής. Η ειδική αυτή έκθεση αξιολογεί το κατά πόσον οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στο παρελθόν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κανόνων δημοσίων συμβάσεων. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στον κύριο Owen Η παρουσίασή του θα ακολουθεί όπως συνήθως με ανταλλαγή απόψεων. Πριν του δώσω το λόγο, να πω ότι έχουμε εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ στην αίθουσα και θα τους δώσω το λόγο προφανώς και για να απαντήσουν σε ερωτήσεις και για να σχολιάσουν την παρουσίαση ε, τον κύριο Αλιάτα, τον κύριο Ζέμπερτ, και τον κύριο Ντεαλμέιδα από την Γενική Διεύθυνση Regio και Grow της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δίνω το λόγο στον κύριο Ον. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να παρουσιάσω την έκθεση αυτή εκ μέρους του Ελεκτικού Συνεδρίου. Την είχαμε ήδη παρουσιάσει στις 15 Οκτωβρίου στην Επιτροπή και στην ΙΜΚΟ τη Δευτέρα την περασμένη. Και μας ικανοποιεί το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο χρόνος που μας δίνεται να εξηγήσουμε. Στην πολιτική λοιπόν της συνοχής έχουμε μια μόνιμη πηγή λαθών αυτό το βλέπουμε σε αιτήσιες εκθέσεις του συνεδρίου εδώ και πολλά χρόνια. Το Κοινοβούλιο ζητά συνεχώς διορθώσεις εδώ και μάλιστα οι αιτήσιες εκθέσεις του συνεδρίου του 2014 που παρουσιάστηκαν ακριβώς την Τρίτη στην Επιτροπή Κόντ στο Κοινοβούλιο έδειξαν ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Έχουμε σοβαρές παραβιάσεις των διατάξεων. Εις 50% περίπου της ε, πρόβλεψης λαθών για την πολιτική συνοχής εντός της περίοδου ελέγχου. Και η μη συμμόρφωση προς διατάξεις των ε, δημοσίων συμβάσεων επηρεάζει ιδιαίτερως την προσθέμενη αξία των συμβάσεων. Θα πρέπει να έχουμε ένα εργαλείο κλειδί για την διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς και της συμμετοχικής ανάπτυξης, όπως και της αποτελεσματικότερης χρήσης των δημοσίων πόρων. Με τον έλεγχο αυτό οικοδομήσαμε επί των πορισμάτων του ελεκτικού συνεδρίου επί τη βάση ακριβώς των ετησίων εκθέσεων. Και το βασικό ερώτημα ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσον η Κομισιόν και τα κρατημέλη λαμβάνουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για να διορθώσουν τα σφάλματα αυτά ή στον τομέα της πολιτικής συνοχή. Επομένως, πολύ σύντομα, πώ διεξήχθη ο έλεγχος αυτός. Συμπεριλαμβανόταν το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξη, το Ταμείο Συνοχή και το Κοινωνικό Ταμείο. Επισκεφθήκαμε τέσσερα κρατημέλη. Την Τσεχική Δημοκρατία, την Ισπανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε κάθε, μία, σε κάθε ένα από τα οποία είχαν ήδη εντοπιστεί λάθη στην περίοδο 2009-2013 σε ελέγχους ε, ε, επιβεβαίωσης και επισκεφτήκαμε επίσης 115 σχετικές αρχές ελέγχου σε 27 συνολικά κρατημέλη και είχαμε και σύντομη έκθεση που απεστάλλει στα ανώτατα όργανα ελέγχου, τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα των κρατών μέλων. Η έκθεση δείχνει ότι και η Κομισιόν και τα κρατημέλη πρέπει να κάνουν περισσότερα για να αντιμετωπίσουν το θέμα. Παραμένουν τα σφάλματα αυτά ή στον τρόπο τον οποίο ε, συνάπτονται οι συμβάσεις επί τη βάση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Συνοχής. Εντοπίστηκαν σφάλματα σε 40% του συνόλου των έργων όπου ελέγξαμε τις δημόσιες συμβάσεις για την ε, περίοδο εκθέσεων 2009 2013 και το 1 τρίτο εξ αυτών σοβαρές παραβιάσεις. 70% των οποίων στο ERDF. Και η ετήσια έκθεση του 2014 δείχνει αντίστοιχη εικόνα. Έχουμε σε 39 από τις 179 ε, είχαμε πολύ σοβαρά, από τις 179 ε, περιπτώσεις που ελέγχθηκαν από την έκθεση, είχαμε πολύ σοβαρές παραβιάσεις. Είχαμε συστημητική ανάλυση των σφαλμάτων, μάλλον ο έλεγχος και η ανάλυση των σφαλμάτων που γίνεται από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη είναι περιορισμένη και δεν υπάρχουν και επαρκή δεδομένα ούτε σε επίπεδο Κομισιόν ούτε σε επίπεδο κρατών μελών. Η Κομισιόν προχώρησε σε μία τέτοια ανάλυση το 2011 χωρίς καμία άλλη επικαιροποίηση έκτοτε. Και ο δείχνει ότι η Κομισιόν και τα κράτη μέλη έχουν ξεκινήσει να αναλαμβάνουν κάποια μέτρα αλλά υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα που μας περιμένει. Η πρόσφατη νομοθεσία μπορεί να καλύψει τα προβλήματα αυτά, αλλά όλα εξαρτώνται από την εφαρμογή. Καταρχάς έχουμε νέες οδηγίες ε, δημοσίων συμβάσεων, όπου ο έλεγχος δείχνει ότι η πιο συστηματική κωδικοποίηση της νομολογίας θα μπορούσε να καλύψει κάποιες από τις παραβιάσεις αυτές, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν από την ακριβώς εφαρμογή από πλευρά των κρατών μελών. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση και τη Δευτέρα εδώ. Συζήτηση επί του θέματος αυτού. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε τους κανονισμούς για τα ευρωπαϊκά διαθωτικά ταμεία οι οποίες όπως γνωρίζετε συμπεριλαμβάνουν αυτές τις προϋποθέσεις εξάντε οι οποίες υποτίθεται ότι εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία και χρήση των απαιτητικών και διαδοτικών ταμείων. Το συνέδριο λοιπόν βρήκε ότι στην αρχή του έτους του 2015 12 κράτη-μέλη δεν είχαν συμμορφωθεί προς τις προϋποθέσεις αυτές, προς το σύνολο αυτών των προϋποθέσεων. Ή στη δημοσιονομική περίοδο την παρούσα, 2014-20. Και στις 15 Οκτωβρίου στην Επιτροπή Κοντ, ευτυχώς τρία από τα 12 αυτά είχαν καλύψει τα σφάλματά τους μέχρι τότε. Βεβαίως δεν μπορούμε να σχολιάσουμε από αυτού. Αλλά μπορούμε να σημειώσουμε ότι εννέα εκ των κρατών αυτών, η Βουλγαρία ή η Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάς, η Κροατία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία. Αυτά τα εννέα κράτη-μέλη, εφόσον ακόμα δεν συμμορφώνονται προς τις προϋποθέσεις δημοσίων συμβάσεων, τότε οι δικές μας συστάσεις ισχύουν. Και αν αυτά δεν εφαρμοστούν μέχρι το ε, τέλος του 2016 θα πρέπει η Κομισιόν να χρησιμοποιήσει την εξουσία της καταλήλως ώστε να διακόψει τις πληρωμές. Οι δράσεις που έχουν αναλυφθεί από την ε, Κομισιόν αρχίζουν σιγά σιγά να στοχοποιούν το σύνολο του προβλήματος με εσωτερική τεχνική ομάδα εργασίας και σχέδιο δράσης που ανακοινώθηκε και αυτά είναι βήματα προς σωστή κατάφυνση αλλά χρειάζεται σωστή ηγεσία ώστε να αρθεί και η πίεση και η ένταση που υπάρχει στα κράτη-μέλη με δύο στόχους. Τη βελτίωση του, των συστημάτων δημοσίων συμβάσεων και την καλύτερη απορρόφηση των αραγικών πόρων. Επίσης σημειώνει η έκθεση ότι τα συστήματα πληροφορικής θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την κατάσταση. Διότι εδώ έχουν μια δυνητική δυνατότητα μετατροπής του τοπίου, αλλά αυτό ποικίλει ανακράτος μέλος. Και η επικαιροποίηση των τραπεζών δεδομένων, όπως η αράκνη τράπεζα δεδομένων της Κομισιόν για την καταπολέμηση της απάτης, ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί πλήρω. ώστε να εξασφαλίσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία. Συνοψίζοντα λοιπόν, το συνέδριο συστήνει τα εξής Πρώτον, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συλλέξουν τα δεδομένα σφαλμάτων ως στη τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των σφαλμάτων αυτών και να τα αξιολογεί στην περιοχή της ε, πολιτικής συνοχής. Δεύτερον, αν οι προϋποθέσεις των διαδικτικών και μεριτικών ταμείων δεν καλυφθούν μέχρι το έτος 16, η Κομισιόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της ώστε να διακόψει τις ε, πληρωμές προς τα κράτη-μέλη που δεν έχουν διορθώσει μέχρι να το πράξουν η Κομισιόν θα πρέπει να επικαιροποιήσει και να δημοσιοποιήσει το εσωτερικό σχέδιο δράσης, να βελτιώσει την ε, ε, διυπηρεσιακή της εσωτερική συνεργασία και να συστήσει μια ομάδα υψηλού επίπεδου για τη βελτίωση της καθοδήγησης. Πέπτον, η Κομισιόν θα πρέπει να διορθώσει, να προχωρήσει μάλλον σε δημοσιονομικές διορθώσεις και να προχωρήσει σε διαδικασίες παραβίασης εκεί όπου ε, απαιτείται υπό τι οδηγίε και έκτον και τελευταίο, η Κομισιόν τα κρατημέλη θα πρέπει να διαρευνήσουν περαιτέρω τις δυνατότητες που παρέχει η... τα συστήματα πληροφορική ή πληροφορική για την συλλογή των δεδομένων και για το data mining. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την εξαιρετική της συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου και με χαρά βλέπουμε ότι συνεφώνησε η Κομισιόν να ακολουθήσει όλες τις συστάσεις μας. Βεβαίως θα το παρακολουθούμε αυτό εμείς προσεκτικά και ελπίζω ότι η έκθεση αυτή θα βοηθήσει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέλη του και ιδιαίτερα την Επιτροπή Ρέτζη για να καλύπτει καλύτερα τα θέματα της ε, πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστώ με στη διάθεσή σας. Thank you. Thank Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Και όλοι μας έχουμε αντίτυπο τη έκθεσης. Έχουμε λοιπόν όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστούμε για την ε, περιεκτική αυτή παρουσίαση. Έχετε λοιπόν το λόγο, συνάδελφοι. Ο κύριος Φαν Νίστελροϊ, για να ξεκινήσουμε με τους ε, Νομίζω ότι όσοι θέλουν να πάρουν το λόγο μπορούν να πάρουν το λόγο, λέει ο κύριος Φαν Νίστελροϊ. Πιστεύω ότι με την ε, παρουσίαση αυτή επιβεβαιώνεται εκ νέου το που σκαλώνει το σύστημα έχοντας ε, διατυπώσει και θέματα σε αιρεσιμότητα εξάντε, αυτό επιβεβαιώνεται ακόμα πιο πολύ. Ερωτώ λοιπόν και εσάς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη στιγμή στην οποία καταλήξατε στο συμπέρασμα για τις χώρες αυτές που δεν πληρούν τα κριτήρια και τη σημερινή στιγμή. Γιατί ουσιαστικά Τώρα ξεκινά την νέα περίοδο. Και μπορεί κανείς να ε, εξετάζει τις διάφορες χώρες αλλά και τις περιφέρειες αναχώρα γιατί υπάρχουν τεράστιες διαφορές ε, μεταξύ των περιφερειών. Στην Ιταλία για παράδειγμα από ό,τι ξέρετε και σε άλλες χώρες. Άρα Κοιτάμε τα κράτη-μέλη, επίπεδο κρατών μελών ή επίπεδο περιφερειακό. Γιατί τελικά ενδεχομένως να στιγματίζουμε ολόκληρες χώρες, όπως στην Ουγγαρία για παράδειγμα, χωρίς να ξέρουμε αυτό τι σημαίνει απαραίτητα. Πείτε μας λοιπόν τι γίνεται, τι διαδικασία ακολουθείτε. Δεύτερη ερώτηση σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκα με επιχειρηματίε από τις κάτω από τη δική μου περιφέρεια. Μας μίλησαν για τις δημόσιες συμβάσεις και την συμμετοχή σε άλλε περιφέρειες στην Ευρώπη. Μα ούτε στο Βέλγιο δεν μπορούμε εμείς να συμμετάσχουμε. Κοιτάμε πως ε, τα τα κονδύλια, πώς πληρούνται οι απαραίτητοι όροι. Πείτε μας όμως γενικά τι γίνεται με τις δημόσιες συμβάσεις. Αν μια Ολλανδική εταιρεία προσπαθεί να πάρει μια σύμβαση στην Ουγγαρία, μπορεί ή δεν μπορεί τελικά. Υπάρχουν προβλήματα, για παράδειγμα, μεταφράσεων και το καθεξής. Μπορείτε λοιπόν να αξιολογήσετε συνολικά τις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρώπη. Κατά πόσον υπάρχει μια τέτοια ανοιχτή αγορά. Κατά πόσον αυτή η αγορά ανθεί. Γιατί βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις να δούμε το σύνολο της ε, πρακτικής εφαρμογής. και θα θέλαμε να ακούσουμε τα, τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τέλη του 2016. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Βον, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο και τον κύριο Φιλ Γουίν για την εξαιρετική παρουσίαση, ως συνήθως. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά ευχάριστα τμήματα στην έκθεση, ιδιαίτερα εκεί πέρα που αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη έχουν πλέον αναλάβει δράση σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη συλλογή δεδομένων. Πρώτο και βασικό σημείο. Χωρί τέτοια δεδομένα, πώ θα τηρηθούν αρχεία, πώ θα αναλυθούν τα προβλήματα στι. Ε, στους δημοσιογεγονισμούς Είναι περίπλοκη η κατάσταση και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συχνά καλούμε τα κράτη-μέλη να, να κοιτάξουν τα θέματα αυτά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, όπου υποτίθεται ότι έχουμε ένα καλό σύστημα ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και εκεί όμως έχουμε προβλήματα, τα οποία δεν παραδεχόμαστε ενδεχομένω δημόσια. Σε πολλές περιφέρειες υπάρχουν προβλήματα με τους νέους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις τις οποίες αναφέρατε στην παρουσίασή σας τώρα. Όταν τα ψηφίσαμε όλα αυτά στο Κοινοβούλιο, θεωρώ ότι ήταν πολλά τα καλά στοιχεία τα οποία περιλαμβανόντουσαν. Περιβαλλοντικές δράσεις των εταιριών, πρακτικά και πρακτικές και αρχεία για την απασχόληση, χρήση τοπικών προμηθευτών. Όλα αυτά ήταν θετικά στοιχεία. Αλλά ότι τελικά τα πράγματα ε, έγιναν πολύ πιο περίπλοκα σε ό,τι αφορά τις ε, δημόσιες συμβάσεις. Ε, μπορείτε λοιπόν να μας κάνετε μια ανάλυση για τους νέους κανόνες αυτούς. Δεύτερο ζήτημα. Αυτός ο ενιαίος έλεγχος σε πολλά μέρη αναφέρεται και μας λένε ότι θα ήθελα ε, να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου επιθεώρησης. Το ελεγκτικό συνέδριο ήταν ε, αντίθετο στο παρελθόν. Και το τελευταίο σημείο το οποίο ήθελα να αναφέρω είναι οι αναστολές και η συλλογή. Το πιο αμφιλεγόμενο τμήμα της παρουσίασης ε, και τη έκθεση, είναι δύσκολο να υπάρχουν αυτόματε αναστολέ και διορθώσει σε πολλά κράτη-μέλη. Τα αντιστατικά ταμεία, για παράδειγμα, ε, χωρούνται σε επίπεδο από το επίπεδο των περιφερειών, των δημοκρατικών και σε κάποιε περιπτώσει και σε πιο χαμηλό επίπεδο. Είναι δύσκολο λοιπόν να πούμε ότι θα υπάρξει ένα αυτόματο σύστημα αναστολή και διόρθωση. Ίσως ενδεχομένω θα έπρεπε να αναζητήσουμε ένα μηχανισμό με κάποια ευελιξία. από πλευρά τη Επιτροπή για να αποφασιστεί κατά πόσον θα προχωρήσει σε διόρθωση και αναστολή. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόμαθιτς, λέει η Πρόεδρος. Αναφέρατε την Κροατία, κύριε Όεν. Η Κροατία γνωρίζω αντιμετωπίζει πολλά ζητήματα σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Η... Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ε, οι δικαιούχοι ε, έχουν εκφράσει παράπονα γιατί πολύ συχνά οι δικαιούχοι ε, ανήκουν στο ίδιο κόμμα με αυτό της κυβέρνησης και πολύ συχνά δεν μπορούν να παραπονεθούν. Ε, δεν έχουν τη δυνατότητα ε, να διαμαρτυρθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την πολύ ξεκάθαρη παρουσίαση. Με εξέπληξε 40% των έργων που εξετάστηκαν ε, πάσχουν από σφάλματα. Εντυπωσιακό. Σχεδόν τα μισά δηλαδή έργα αντιμετωπίζουν τέτοιου είδου προβλήματα. Δεν συμμορφώνονται με τους ίδιους κανόνες που τα διέπουν. Οπότε η ερώτηση είναι η εξή. Γνωρίζω από την προσωπική μου ε, εμπειρία στην Ολλανδία ότι ο κανονιστικός υπερθεματισμός είναι και αυτός ένα πρόβλημα. Πολύ συχνά σε εθνικό επίπεδο οι κανόνες είναι πιο αυστηροί από ότι η αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Λάβατε υπόψη και τους εθνικούς και περιφερειακούς κανόνες για, τους, για τις δημόσιες συμβάσεις. Ε, αποτελούν αυτοί οι κανόνες τμήμα των ε, αριθμητικών στοιχείων που μας δώσατε ή εξετάσετε μόνο τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αυτό, αυτό το ποσοστό σφάλματος αφορά τη συμμόρφωση μόνο με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ή και με τους εθνικούς και περιφερειακούς κανόνες. Φανταστείτε να λάβουμε υπόψη και τους ε, ε ειδικού ε, τοπικούς κανόνες, αν δεν τους έχετε λάβει. Το ποσοστό σφάλματος θα ήταν ακόμα υψηλότερο. Θα πρέπει να πάρουμε πολύ στα σοβαρά τις συστάσεις. Νομίζω ότι οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για, τους, ε, για τις δημόσιες συμβάσεις ε, όταν δεν λαμβάνονται υπόψη από χώρε όπως αυτές που αναφέρετε θα πρέπει αυτή η κατάσταση να οδηγεί σε δημοσιονομικές διορθώσεις και κυρώσεις. Γιατί, Γιατί θα πρέπει να είμαστε συνεπείς ε, με αυτά που έχουμε αποφασίσει στο παρελθόν. Είναι μια πολύ υγιής, πολύ λογική σύσταση. Να λάβουμε δράση εκεί που πρέπει. Ευχαριστώ κύριο Σόμερτζέ. Κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση αυτή. Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτον, πιστεύετε ότι σε αυτές τις δαπάνες για τις δημόσιες προμήθειες υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά την, ε, ε, ε κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με συγκεκριμένους τομείς όπως για παράδειγμα ο, οι αγροτικές επιδοτήσεις. Ε, δεύτερον, σε ό,τι αφορά το ποσοστό σφάλματος που αναφέρατε, θα μπορούσατε να μας πείτε σε αυτό το ποσοστό τι αντιστοιχεί σε απάτη και διαφθορά. Ποιο τμήμα αυτού του ποσοστού. Επίσης, έχετε στοιχεία για το 2014. Τρίτη ερώτηση. Ποια, είναι η δράση της Όλαφ, της Πίσης κατά πολέμησης απάτης, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Λειτουργεί καλά η Όλαφ ή πιστεύετε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θέμα που ήδη συζητείτε. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα μείωνε την απάτη και τη διαφθορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Βάνα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, παρουσιάσεις αυτές ε, και τις εξηγήσει. Νομίζω ότι οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να μειωθεί το ποσοστό σφαλμάτων. Και όπως επιστώνουμε από πολλές δημοσιεύσει. είναι αρκετά σαφές ότι η βασική αιτία δεν είναι ε, η απάτη, η διαφθορά, αλλά τα ελλείμματα στις διοικητικές ικανότητες, τα σφάλματα, τα απλά σφάλματα. Άρα θεωρώ ότι χρειάζεται capacity building, ανάπτυξη δυναμικού ε, και αύξηση, αν θέλετε, της αποπτικότητας για να μειωθεί το ποσοστό σφαλμάτων. Ένα άλλο θέμα που θα με ενδιέφερε. Η Γενική Διεύθυνση Ρέτζη και η Διεθνή Διαφάνεια έχουν προτείνει ένα πακέτο για την ακαιρεότητα, integrity package για κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές κατά των απατών, της διαφθοράς, των εκβιασμών και άλλων τέτοιων πρακτικών. Και συνοδεύεται αυτό το πακέτο και από ένα σύστημα παρακολούθησης. Κάποια έχουν ακολουθήσει αυτό το εργαλείο. Πιστεύετε είναι ενδεδειγμένο αυτό το μέσο για τη μείωση των σφαλμάτων στα κρατη και μία δεύτερη ερώτηση για την ε, χρήση, την εφαρμογή της αρχής ε, του καλύτερου παρόχου κατά τις αρχές του φθηνότερου παρόχου. Σήμερα που μιλάμε για την καλύτερη χρήση των ε, χρημάτων του φορολογούμενου, θα πρέπει να έχουμε υπόψη και την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα του αποτελέσματος. Άρα να είναι ο καλύτερος αυτός που επιλέγεται, όχι ο φθηνότερος. Από πλευράς της Αυστρίας, η μικρή δήμη αντιμετωπίζουν προβλήματα αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν ακριβώς αυτή την αρχή του καλύτερου παρόχου ε, ε, γιατί πολύ απλά είναι ανέφικτο αυτό, δεν ε, μπορούν να το δικαιολογήσουν. Κατά πόσο λοιπόν θα μπορούσαμε να προωθήσουμε αυτό το πακέτο θα ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντεμάτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση η οποία είναι ανησυχητική αλλά αποτυπώνει την πραγματικότητα εμείς που βρισκόμαστε στο πεδίο τα γνωρίζαμε αυτά. Βεβαίως το να βλέπει κανείς τα υψηλά αυτά ποσοστά μας κινητοποιεί ακόμα περισσότερο να απαιτούμε από την Κομισιόν να λάβει μέτρα. Τώρα η ερώτηση μου είναι αν μπορείτε να μας πείτε <clears throat> ποιες κατηγορίες φαλμάτων υπάρχουν ήδη και αν διαφέρουν χώρα ή ανά περιφέρεια Και μήπως τελικά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου είναι αυτά που ε, συγκεντρώνουν τα περισσότερα προβλήματα. Επίσης, αυτά τα σφάλματα θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι εξαρτώνται από ελλειπή ειδίκευση ή αποτελεσματικότητα των εθνόντων ή είναι το ίδιο το σύστημα που ενέχει προβλήματα. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Ολμπρέχτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είχαμε το χρόνο να διαβάσουμε το σύνολο του κειμένου, βεβαίως. Ίσως να συζητήθηκε σε άλλες επιτροπές, αλλά το... η ερώτησή μου είναι το πρόβλημα είναι πού. Ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν ένα σύστημα που να προσαρμόζεται καλά προς τις οδηγίες. Δηλαδή δεν είναι προετοιμασμένα για την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή έχουν την κατάλληλη νομοθεσία τα κράτη-μέλη αλλά δεν την ακολουθούν. Και επομένως γίνονται αυτά τα σφάλματα. Δηλαδή η ερώτηση είναι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία τι γίνεται. Είναι εκείνη επαρκώς σαφής για τα κρατημέλη και για την σωστή εφαρμογή της. Αν θέλουμε να διορθώσουμε τα σφάλματα ε, πρέπει να δούμε πού βρίσκονται εμπόδια, πού συγκεντρώνονται τα σφάλματα, τι είδη σφαλμάτων, τι τυπολογίες. Δηλαδή κατά την άποψή σας, πού εστιάζεται το πρόβλημα. Διότι αν δεν έχουν την απαραίτητη νομοθεσία τα κράτη-μέλη, θα υποστούν τις κυρώσεις. Αν οι τελικοί δικαιούχοι δεν ακολουθούν τους κανόνες. Είναι οι κανόνες που είναι ασαφείς ή αυτοί έχουν κάνει κάποιο λάθος. Και ποιος πρέπει τελικά να υποστεί κυρώσεις. Η κυρία Μπρέσο λέει πρόεδρος, ευχαριστώ πρόεδρε. Λέει η κυρία Μπρέσο. Εγώ ήθελα να καταλάβω καλύτερα αυτό που εννοείται όταν λέτε κωδικοποίηση των σφαλμάτων γιατί όπως ανέφερε και ο κύριος Βον, εγώ είμαι εισηγήτρια για κάποια θεσμικά ζητήματα και το θίγω το θέμα αυτό. Και κατά την άποψή μου είναι απαραίτητο να, αν θέλετε, να καταλογοποιήσουμε τα σφάλματα ώστε να διακρίνουμε την απάτη από το σφάλμα. Δηλαδή την πρόθεση να εξαπατήσουμε ή τα σφάλματα που απορρέουν από κενά της νομοθεσίας ή από κενά συστημικά ή συστηματικά που θα μπορούσαμε να τα επιδιορθώσουμε εφόσον κατανοούσαμε καλύτερα που βρίσκονται. Άρα λοιπόν αυτή η διάκριση είναι πολύ σημαντική κατά την άποψή μου γιατί θα γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε μια διαθεσμική συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία που λέμε και την διαφανέστερη και καλό θα ήταν να διακρίνουμε το σβάλμα από την απάτη ή την παραβίαση. Γιατί μέσα στην όλη ασάφεια ίσως αυτή η διάκριση κάπως χάνεται. Και θα ήθελα να το καταλάβω καλύτερα, διότι συμφωνώ απολύτως ότι είναι απόλυτη η ανάγκη να δούμε τις κατηγορίες και τις τυπολογίες των σφαλμάτων προκειμένου να νομοθετήσουμε διαφορετικά είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό ακόμα επίπεδο αν το σφάλμα προέρχεται από μας για να το πω έτσι. Αυτή η διάκριση λοιπόν είναι πολύ σημαντική όπως και η άλλη τα μεγάλα κράτη έχουν περιφερειοποιήσει την πολιτική συνοχή. Και επομένω πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη διάκριση των ευθυνών μεταξύ των διάφορων, ε, των διάφορων δημοσίων φορέων. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλουμε να καταλάβουμε ποιος σφάλει χωρίς να επιβάλλουμε κυρώσεις πάνω σε εκείνους που δεν έχουν σφάλει. η νομοθεσία για τη δημόσια συμβάσεις ε, σχεδόν παντού είναι θέμα που εμπίπτει εν πάση σε αρμοδίες των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μάλκοβα για την επόμενη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω λοιπόν ότι πρόκειται να... Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε και νομίζω ότι αν υπάρχουν σφάλματα θα πρέπει να αναφέρονται οι πληρωμέ. Αυτό θα ήταν ασφαλώ πάρα πολύ απλό τρόπο αντιμετώπιση, αλλά αυτό θα πρέπει να αποτελεί και την τελευταία λύση. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Έχουν ληφθεί μέτρα στην Επιτροπή των Περιφερειών. Γιατί αν μία χώρα δεν πληρεί την αιρεσιμότητα εξάντια, αυτό θα επηρεάσει ασφαλώς και τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, τις μειονεκτούσες ε, περιοχές. Ως εκ τούτου. Διαπιστώνουμε ότι αυτό ισχύει από τα στοιχεία που μας παρουσιάζει η έκθεση. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με την Επιτροπή των Περιφέρειων, να μιλήσουμε και με τις κατοχώρες και με την Σλοβακία που θα προετρέψουν του χρόνου. Να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν στο θέμα αυτό και στα πλαίσια της Επιτροπής μας και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τις αιτίε των σφαλμάτων. Εγώ υποθέτω ότι το μεγαλύτερο τμήμα των ε, σφαλμάτων δεν είναι ειστερημένα. Του χρόνου λοιπόν στην αξιολόγηση ελπίζω να έχουν διορθωθεί αυτά τα σφάλματα και πιστεύω λοιπόν ότι από κοινού με την Επιτροπή των Περιφερειών και με τις ε, χώρες ε, οι οποίες θα προεδρεύσουν θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Μάλιστα, θέλετε να πάρετε και στο λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να αδράξω την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον ομιλητή για την έκθεση. Πολλά ζητήματα θίγονται αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Και θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Δεν πιστεύετε ότι υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα στον τομέα αυτό. Το γεγονό δηλαδή ότι το σύστημα δημοσίων συμβάσεων είναι τόσο περίπλοκο, τόσο πολυσύνθετο. Υπάρχουν οι οδηγίε, υπάρχουν και διάφορε καταστάσει όπου κάποια κάτι μέλη αποφασίζουν ένα κανονιστικό υπερστατισμό και ύστερα υπάρχουν και καταστάσεις όπως αυτές που έδειξε ο κύριος Όλμπρεχτ, όπου κάποιες, ε, κράτε, από κάποιες ε, χώρες δεν εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία. Και τελικά η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται είναι η εξή. Α υποθέσουμε ότι είμαστε δικαιούχοι. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα λαβύρινθο πραγματικό ε, νομοθεσιών και κανονισμών είναι αδύνατο να μην διαπράξουμε σφάλματα, όχι θελημένα. Ανεξάρτητα λοιπόν από τις συστάσεις που μας παρουσίασε το ελεκτικό συνέδριο, οι οποίες ασφαλώς και έχουν την αξία τους. Μήπως όμως το πρώτο βήμα θα έπρεπε να είναι η απλοποίηση, η απλούστευση, μήπως αυτό το μήνυμα θα έπρεπε να αποστείλουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να δώσει αυτό το έναυσμα, αυτό το κίνητρο και προς τα κράτη-μέλη Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Πότσακ θέλει να θέσει και αυτό ένα ερώτημα. Mm, Θα ήθελα να δώσω μια συνέχεια στο ερώτημα του συναδέλφου Χέντμαν στο σημείο 33 της έκθεσης. Αναφέρεται ότι ορισμένες ε, χώρες αναφέρουν μόνο ελάχιστο αριθμό παρατυπιών στην Όλαφ στην Ισπανία από το 2007 μέχρι το 2013 για παράδειγμα ε, δεν αναφέρθηκε καμία παρατυπία που να συνδέεται με απάτη. Κάτι που είναι τουλάχιστον παράξενο. Το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί αυτά τα στοιχεία ως αληθοφανή, ότι δηλαδή πραγματικά δεν γίνονται απάτες, σε αυτές τις χώρες γιατί πραγματικά θα ήταν εξαιρετικό αν συνέβαινε αυτό. Στο σημείο 29 που αφορά την τσεχική δημοκρατία αναφέρεται ότι πολλές αρχές δίνουν διαφορετικές νομικές ερμηνείες για τα ίδια πράγματα. Πώς θα αντιμετωπίζετε κάτι τέτοιο στο ηλεκτρικό συνέδριο. Ποια από τις ερμηνείες γίνεται δεκτή. Ευχαριστώ. Ο κ. Ρος, τελευταίος ομιλητής. Κ. Ράους. Ε, δεν θα πω πολλά διότι τα περισσότερα πόσα ήθελα να πω έχουν ήδη λεχθεί και ερωτηθεί. Να ε, ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Όουεν για την σαφήνεια της παρατήρησης της ε, παρουσίασής του και να πω πόσο σημαντικές είναι τέτοιου είδους εκθέσεις. Το πανόραμα είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο. Είναι ανησυχητικό. Ασφαλώς θα πρέπει να απλοποιήσουμε τους κανόνες, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να είμαστε πολύ απαιτητικοί σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης. Η πολιτική συνοχής είναι πάρα πολύ σημαντική για να αντιμετωπίζουμε σενάρια όπως αυτά που μας παρουσίασε σήμερα ο κ. Σόβεν. Και τα πιο φτωχά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα θα πρέπει να κάνουν προσπάθεια να συμμορφωθούν γιατί έτσι θα ωφεληθούν όλοι. Thank you. Thank you very much. So we finalized this round. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι ολοκληρώθηκαν ε, οι ερωτήσει των μελών της Επιτροπής Ρέτζη. Βλέπετε ότι είναι πολύ άριθμες και κάποιες εξ αυτών είναι στον τομέα αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά θα δώσω πρώτα το λόγο σε εσά, κύριε Ουμ, και μετά στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσουν τις ερωτήσεις αυτές. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για το έντονο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι 13 μέλη της Επιτροπής είναι εδώ, τουλάχιστον, και πραγματικά σας συγχαίρω. Είναι αριθμός ρεκόρ αυτός. Δεν είμαι βέβαιο ότι θα απαντήσω σε όλε τι ερωτήσει σα, αλλά μην στάσετε να με ξαναρωτήσετε. Μα ρωτήσατε για τα κράτη-μέλη, κύριε Φανίστε Ρόι, και για τι περιφέρειε. Ναι, κοιτάξτε, τουλάχιστον 12, 13, 15 ενδεχομένω στην Ουαλία. Θεωρούμε ότι το 15 είναι τυπικό αριθμό πάντα. Κύριε Φανίστε Ρόι, για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σα. κατά πόσο τα προβλήματα εστιάζονται στα κράτη-μέλη ή σε επίπεδο περιφερειών. Και τα δύο. Υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα από τα τέσσερα κράτη-μέλη τα οποία εξετάσαμε. Κοιτάξαμε ασφαλώς και εξετάσαμε τρία μεγάλα κράτη-μέλη με μεγάλο ιστορικό, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και δυστυχώς βλέπουμε ότι έχουν μεγάλο ποσοστό σφάλματων. Είναι διαφορετικά τα συστήματα της διοίκηση, αλλά κάποιε από τι πρακτικέ ήταν ευρέω δεδομένε. Δεν κάναμε ανάλυση τέτοια για να δούμε κατά πόσο να υπήρχε πρόβλημα ε, σε συγκεκριμένε περιφερειέ. γιατί αυτό ως στατιστικό δείγμα δεν είναι ε, αξιόπιστο. Αλλά ένα θέμα είναι να κατανοήσουμε το επίπεδο στο οποίο εστιάζονται και από το οποίο προκύπτουν τα σφάλματα. Ένα πρόβλημα το οποίο και σημειώσαμε ήταν το εξή και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση. Είναι το θέμα τη συνδεσιμότητα τη μεγάλες αυτέ χώρες μεταξύ τη κεντρική κυβέρνηση και τη τοπική αυτοδιοίκηση. Και έτσι λοιπόν είδαμε μία σειρά εξαιρετικών πρωτοβουλειών που αναλαμβάνονται σε επίπεδο κεντρική κυβέρνηση για σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την κεντρική διαμόρφωση διαγωνισμών ή στην Ιταλία για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αλλά ο βαθμός στον οποίο αυτή η πρωτοβουλία έφτανε και στις περιφέρειες ε, αποτελεί ένα πρόβλημα σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα. Ελπίζω να υπάρξει μεγαλύτερη κίνηση και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την πάροδο του χρόνου. Ο κύριος Βον, σας ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας και για τις παρατηρήσεις και για το γεγονός ότι ακούσατε δύο φορέ την, την ε, παρουσίασή μου. Κάποια καθημερι όντως αρχίζουν και κινητοποιούνται. Αυτό είναι καλό. Αναφέρατε ότι και στη χώρα μας ε, υπάρχουν προβλήματα και η φετινή έκθεση καταδεικνύει ότι υπάρχουν σοβαρά ασφάλματα. Θα μιλήσουμε για την αιτήσια αυτή έκθεση στο Λονδίνο σε ανώτερους αξιωματούχους συμπεριλαμβανομένων και αξιωματούχων από την Βορεια Ιρλανδία, τη Σκοτία, την Ουαλία για να αντιμετωπίσουμε την πηγή των προβλημάτων γιατί κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να βελτιωθεί. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τα ίδια προβλήματα ή του ίδιου τύπου προβλήματα σε όλες τις χώρες. Είναι οι κανόνες τώρα για τις δημόσιες προμήθειες. Περιλαμβάνουν κάποια θετικά στοιχεία υπήρξε μια διάθεση απλούστασης, απλοποίησης, προκειμένου να υπάρχει ισορροπία στην εφαρμογή. Η περιβαλλοντική και η κοινωνική πτυχή. Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο καλώς όρισε ιδιαίτερα στο Κοινοβούλιο, αλλά προφανώς οι νέοι κανόνες συνεπάγονται και νέες περιόδους ε, προσαρμογή σε μεταβατικές περιόδους όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για ασφάλματα. αλλά η γενικότερη κατεύθυνση των νέων κανόνων είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια, μεγαλύτερη απλούστευση και νομίζω ότι αυτό είναι πρόσδεκτο. Αυτή η απλούσταση είναι κάτι το οποίο το ελεγκτικό συνέδριο εδώ και χρόνια ζητά, αλλά η εφαρμογή, η διαδικασία εφαρμογής από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα σχολιαστεί μάλλον ως κάτι το πιο περίπλοκο. Ένας ενιαίος έλεγχος, μία ενιαία επιθεωρήση θα βοηθούσε. Όπως ξέρετε, το ελεγκτικό συνέδριο εξακολουθεί να ανακαλύπτει σφάλματα τα οποία θα έπρεπε να έχει ανακαλύψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα σε, σε βάθος χρόνου θα πρέπει να βρεθεί ένα σύστημα επιθεώρησης ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κινηθούμε προ την κατεύθυνση αυτή. Προς το παρόν όμως επιτελούμε τα καθήκοντα τα οποία μα έχει αναθέσει η συνθήκη για την αναστολή και τι διορθώσει. όπω είπε και η συνάδελφό σα, είναι δύσκολο να υπάρχει αυτοματισμό και προφανώ είναι συντεκτική ευχαίρεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πώ θα ερμηνεύσει θέματα κριτηρίων ερεσιμότητα εξάντε. Οι κανονισμοί όμω είναι αρκετά ξεκάθαροι πιστεύω και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αποφασισμένη ότι αν μέχρι το 2016 κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν πληρούνται οι όροι εξάμπτε αιρεσιμότητα, θα πρέπει να υπάρξει αναστολή. Τώρα, το τι θα σημαίνει αναστολή αυτή, σε τι κονδύλια θα αναφέρεται, σε ποιου τομεί κλπ. αυτό είναι κάτι άλλο θα πρέπει αναλογικά να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως θεωρεί ότι αρμόζει. Αλλά νομίζω ότι είναι σαφείς οι κανόνες σε ό,τι αφορά τους όρους εξάντε και αν δεν πληρούνται μέχρι το τέλη του 2016. Έχουμε όμως ένα χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Και σημειώνουμε το πρόοδος, όπως σας είπα, από κάποια κρατημέλη για την κυρία Τόμας κατά πόσον υπάρχει ένα σώμα για την υποβολή ενστάσεων από πλευρά των δικαιούχων. Δεν ξέρω τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι σε κάθε κράτο μέλος πλέον υπάρχει ένα ανώτατο ελεγκτικό όργανο και νομίζω ότι υπάρχει μία αύξηση των ενστάσεων και μία, θέλετε, αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών υπάρχουν και οι διαμεσολαβητές, διαμεσολαβήτριες οι οποίες μπορούν να εισακούσουν αυτές τις ενστάσεις και τις προσφυγές. Αλλά σε αυτό καλύτερα να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Φαμίλτεμπερ. Για το κατά πόσο ο υπερθεματισμός ο κανονιστικός αποτελεί ένα ζήτημα. Ναι, Το απιστώσαμε αυτό, για παράδειγμα, η Τσεχική Δημοκρατία με τι καλύτερε προθέσει έκανε πιο πολλά για να εφαρμόσει τη δημοθεσία. Υπάρχει και θέμα διαφορετική ερμηνεία των οδηγιών. Αυτό το επισημαίνουμε στην σελίδα 29α και β σε ό,τι αφορά την Ιταλική ερμηνεία για την ε, ερμηνεία, διαφορετική ερμηνεία των συμβάσεων και ο κ. Ανέση ρώτησε κατά πόσον υπάρχουν προβλήματα και σε άλλους ε, τομείς ε, της πολιτικής όπως η ΚΑΠ. Εμείς εστιαζόμαστε, ναι, μεν, αλλά εμείς εστιαζόμαστε στα ταμεία συνοχής ε, και γίνεται μια παράλληλη έρευνα για τα αγροτικά θέματα. Είναι πολύ παρόμοια τα αποτελέσματα. Εμείς εστιαζόμαστε στην συνοχή γιατί εκεί είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά ασφαλμάτων σε τέτοιου μεγάλους τομείς ε, δαπάνης κοντιλίων. Ανάλογες όμως και είναι και κατάσταση και στη και στη Γεωργία. Τώρα, σε δύο φάρτα ποσοστά απάτης, δίνουμε κάποια αριθμητικά στοιχεία για το 2015-2016, ως 6, συγγνώμη. Δεν έχω άποψη για το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όχι. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών να το αποφασίσουν. Το ίδιο ισχύει και για την απάντησή μου για το κατά πόσο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πακέτο, αυτό το σύμφωνο διαφάνειας. Δεν ξέρω. Εμείς εδώ και χρόνια ζητούμε μεγαλύτερη διαφάνεια και η γνωμοδότηση που δημοσίευσαμε πέρυσι για την ε, πρώτη ετήσια έκθεση απάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι και έλεγε ότι χρειαζόμαστε πιο πολλά δεδομένα για μεγαλύτερη διαφάνεια. Άρα στο πνεύμα αυτό πρέπει να πω ότι είναι σύμφωνο για την κυρία Νταμάτα τώρα. Δεν κάνουμε ανάλυση των σφαλμάτων αναπεριφέρεια όπως σας είπα, αλλά δώσαμε όσο πιο πολλές πληροφορίες γίνεται, ιδιαίτερα στα παραθύματα 1 και 2 για το είδος, τον τύπο των σφαλμάτων και κάναμε και μία ανάλυση σε ό,τι αφορά τα σοβαρά και μη σοβαρά σφάλματα. Τα σοβαρά σφάλματα, για να είμαι σαφής, είναι τα σφάλματα όπου θεωρούμε ότι επιλέχθηκε λάθος πάροχος για την σύμβαση. Είναι σοβαρό αυτό το λάθος και δεν τηρείται η αρχή της ε, καλύτερης της επιλογής που έγινε τα προβλήματα, κύριε Ολμπρέχτ. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα μοναδικό πρόβλημα, μια μοναδική αιτία. Η έλλειψη διοικητικής ικανότητας, ο ανεπαρκής σχεδιασμός, αυτά αποτελούν μεγάλα ζητήματα και συμφωνώ ότι πολλοί φορεί διαμαρτύρονται για την μεγάλη περιπλοκότητα. Και αυτό το αντιμετωπίζουμε στην οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό είναι σημαντικό. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι καλή μεταφορά της οδηγίας, δεν είναι σωστή η ερμηνεία της οδηγίας σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν επιπροσθετοί κανονισμοί. Και θεωρούμε ότι ναι, και η απάτη μπορεί να αποτελέσει αιτία για τα σπάλματα αυτά. Αν και είναι δύσκολο να το αποδείξουμε αυτό, η κυρία Μπρέσο, κατά πόσον η κωδικοποίηση, η καλύτερη κωδικοποίηση των σπάλματων θα μας βοηθούσε και κατά πόσον θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε ποια σπάλματα οφείλονται σε απάτη και σε, ποια, σε ποιες περιπτώσεις το θέμα είναι απλά η περιπλοκότητα της νομοθεσίας. Όπως σας είπα, αν υπάρχει καταφανής απάτη, παρέχουμε τα στοιχεία αυτά άμεσα στην Όλαφ. Στον πίνακα 1 στην ε, σελίδα 18 υπάρχει μια αναφορά των σοβαρών και των ε, ίσονων σφαλμάτων. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ε, βοηθητικό, ό,τι πιο διευκρινιστικό μπορέσαμε να σας παρέχουμε σε ό,τι αφορά σφάλματα. Το κατά πόσο για πάτη ή όχι, αυτό θα το καθορίσουν άλλοι. Κυρία Ζωνκόβα. για το θέμα του αυτοματισμού. Υπάρχει ένας αυτοματισμός για την περίπτωση που δεν θα πληρούνται οι όροι για την εξάντερεσιμότητα, αλλά υπάρχει και μια διακριτική ευχαίρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν και πολλά επικοδομητικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη όπου αντιμετωπίζουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα και χαίρομαι να σας πω που μας, ε, ότι μας κάλεσαν σε μια κοινή συνάντηση μεταξύ της Επιτρόπου Κρέτσου και Πέσκα για τη συνεργασία μεταξύ των επιτρόπων αυτών. Και χαίρομαι πολύ λοιπόν που 1η Δεκεμβρίου θα έχουμε συνάντηση για την ατζέντα αυτή. Ο κ. Χέτμαν, κατά πόσον υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ε, η περιπλοκότητα και το Ευρωπαϊκό το Ελευθερικό Συνέδριο ζητά απλούστευση εδώ και χρόνια. Και σε ό,τι αφορά θέματα εφαρμογή. Εδώ μπορεί να θέλει να σχολιάσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Πότσερ. δεν μπορούμε να πούμε κάτι πέρα από αυτά που είπαμε στην έκθεσή μας. Είμαστε περίεργοι που κάποιες ε, χώρες στις εκθέσεις τους ε, προς την Όλαφ δεν επισημαίνουν τις υποθέσεις όπου έχει εντοπιστεί απάτη. Δεν είναι μόνο μία αυτή χώρα, αρκετές το κάνουν. Ενδεχομένω να έχει να κάνει με την απροθυμία να επισημανθούν ω περιπτώσει απάτης, κάποιες περιπτώσει και κάποια φάλματα τα οποία δεν έχουν αποδειχθεί ότι αφορούν απάτη. Και βλέπουμε για παράδειγμα στην Ισπανία ε, οι εισαγγελικές αρχές ε, αναφέρονται και στον τύπο ότι έρευνουν τα χειροτήματα. Τέλος, ο κύριος Ρούες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια που κάνετε και πιστεύω ότι συμφωνήσατε μαζί μας ότι ε, αν υπάρχουν κανόνες και νόμοι και κανονισμοί θα πρέπει να τηρούνται. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Αυτό είναι ουσιώδες για ένα κοινοβούλιο, είναι και ουσιώδες για το ρόλο του ελεγκτή και νομίζω ότι με αυτή την νότα μπορούμε να κλείσουμε όπως αρμόζει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις λεπτομερείς απαντήσεις. Θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Λιάτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε τρεις από την Κομισιόν εδώ. Οπότε εγώ θα κάνω κάποια σχόλια και μετά ο Διευθυντής ε, ελέγχου και η Διευθύντρια της, των Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Growth θα συμπληρώσουν. Τρία σχόλια έχω να κάνω εγώ ίδια. Πρώτον, συμμεριζόμαστε και οι τρεις μας και γενικότερα η Κομισιόν τους, τον τελικό στόχο. Ο στόχος είναι η αποτελεσματική εφαρμογή των κανονών δημοσίων συμβάσεων ε, στο πλαίσιο των διαστολικών ταμείων. Και αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιλέγουν τα καλύτερα έργα στην καλύτερη τιμή. Και όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Θέλουμε δηλαδή να ε, βλέπουμε περισσότερες δημοπρατήσεις διασυνοριακές. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη που έχουν σοβαρά σχέδια καταπολέμησης της ε, διαφθοράς ή αποφυγής της όλης διαφοράς στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις συστάσεις της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Owen για τη δουλειά του, για την συνεργασία που είχαμε μαζί του στο παρελθόν δεχόμαστε όλες τις συστάσεις του και θα τις εφαρμόσουμε. Δεν θα σχολιάσω όλες τις συστάσεις προφανώς. Ε, μερικά σημεία μόνο. Ευχαριστούμε πολύ για την σύσταση που αναφέρει ότι το πρόγραμμα δράσης της Κομισιόν για τη βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων δημόσιας δημοσίων συμβάσεων από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να περάσει σε υψηλότερο πέδο, να υιοθετηθεί σε πέδο επιτρόπου. Η κυρία Κρέτσου και η κυρία Μπιενκόφσκα θα συναντηθούν στις 2 Δεκεμβρίου με τον κύριο Όουεν για πρώτη φορά έτσι ώστε πραγματικά να εγκρίνουν αυτό το πρόγραμμα δράσης και να αρχίσει η παρακολούθηση της εφαρμογής του. Θα ακολουθήσουν τακτικές συνεδριάσεις στο πλαίσιο της εφαρμογή του προγραμματό δράση. Τρίτον, η τρίτη μου παρατήρηση, να δώσω ορισμένα παραδείγματα της προσέγγισης μας σχετικά με την σύνδρομη που δίδουμε στα κράτη-μέλη προκειμένου να βοηθήσουν να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους. Έχουμε προληπτικά εκ των προτέρων μέτρα ε, και διορθωτικά μέτρα. Εγώ θα μιλώσω για τα πρώτα, οι συνάλφοι για τα δεύτερα. Σε ό,τι αφορά την πρόληψη, ε, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τη Γενική διάθεση GROW γιατί έχουμε κοινούς στόχους. Μαζί αναπτύξαμε μερικά εθνικά προγράμματα δράσης, ιδιαίτερα στις χώρες οι οποίες αναφέρονται ως χώρες που δεν πληρούν τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες. Εν τω μεταξύ βέβαια, ε, τρεις χώρες από αυτές που ανέφερε ο κ. Σόουεν συμμορφώθηκαν και εφάρμοσαν τις δράσεις που έπρεπε. Οπότε θεωρούμε ότι συμμορφώνονται πλήρω η Μάλτα, η Πολωνία και η Λετωνία συγκεκριμένα. Για τις υπόλοιπες χώρες έχουμε εθνικά προγράμματα δράσης με δράσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν πριν το τέλος του 2016. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα γιατί ακούσαμε και συγκεκριμένε ερωτήσεις. Ζητούμε να κωδικοποιηθεί επαρκώς η νομοθεσία. Δηλαδή η νομοθεσία να μην είναι μοιρασμένη σε διάφορα κείμενα ε, απροσπέλαστα. Θέλουμε ε, να κωδικοποιηθεί και αυτό ζητάμε από αυτά τα κράτη-μέλη. Επίσης δίνουμε πολύ έμφαση στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης γιατί είναι σημαντικό οι, αυτοί που δημοπρατούν και σχετίζονται με δημοπρατήσεις να είναι πραγματικοί επαγγελματίες. Ε, Επίσης δίνουμε μεγάλη σημασία τα κατάλληλα εργαλεία που θα βοηθήσουν ε, στην αποφυγή εισφαλμάτων, εγχειρίδια και άλλου τύπου υλικό που θα καθοδηγεί τους επαγγελματίες αυτούς στη δουλειά τους. Μετά, έχουμε και ένα πιλωτικό πρόγραμμα μαζί με την ε, Διεθνή Διαφάνεια ε, για τη δημιουργία πακέτων ε, ε, συμφωνιών μεταξύ διεθνών κυβερνητικών οργανώσεων για τη διαφάνεια και από την άλλη πλευρά εθνικών αρχών έτσι ώστε ε, να αποφεύγονται πράξεις που έχουν σχέση με τη διαφθορά. Το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα θα λάβει η χώρα το 2016, θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα και θα δούμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε και να γενικεύσουμε αυτή την εμπειρία της, των συμφώνιων ακαιρεότητας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, εκ των προτέρων ρεσιμότητες, όταν, την πρώτη, όταν κάναμε την πρώτη αξιολόγηση, ε, την κάναμε σε εθνικό επίπεδο, αλλά ιδιαίτερα σε μεγάλες χώρες όπου υπάρχουν πολλές περιφέρειες και διαφορετικές μεταξύ τους, τελικά στο τέλος του 2016 η ανάλυση που θα γίνει σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση θα γίνει και σε επίπεδο περιφερειακών προγραμμάτων, εκεί που υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα. Αν σε ορισμένες περιφέρειες έχουν, ε, αν ορισμένες περιφέρειες έχουν συμμορφωθεί και άλλες όχι, παρόλο που η χώρα δεν συμμορφώνεται στο σύνολό της, θα αποφύγουμε δημοσιονομικές διορθώσεις και κυρώσεις στις περιφέρειες οι οποίες συμμορφώνονται. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους μου αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ ο κ. Ζέλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Από το τμήμα Audit ε, της ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ ΡΕΓΚΙΟ. θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Όουνεν και την ομάδα του για όλη τη δουλειά που έκαναν ε, στις δημόσιες συμβάσεις. Είναι αλήθεια και λέγεται στην έκθεση ότι αυτό δεν είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πολιτικής συνοχής. Ωστόσο, είναι μία από τις βασικές ε, συνθήκες και όρους υπό τις οποίες ε, εφαρμόζουμε τα προγράμματά μας και το συνέδριο εξηγεί γιατί η συχνότητα είναι αυξημένη στα προγράμματα της ΓΔ Εμείς έχουμε προχωρήσει σε πάρα πολλούς ελέγχους ε, τα τελευταία δύο χρόνια και περισσότερο με κατευθύνσεις ε, κατάρτιση, συστάσεις κατάρτισης προς τα κάτι μέλη κτλ. Το σχέδιο δράσης εξηγείται η εμφάνισή του δηλαδή τώρα, διότι έχουμε διευρύνει τις δράσεις και τις αρμοδιότητες για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλα τα επίπεδα. Τώρα σχετικά με τα σφάλματα και τα κενά που θίγει η έκθεση, που καταλήγουν σε σημαντικές ε, δημοσιονομικές επιπτώσεις και διορθώσεις, οι δράσεις που πρέπει να αναλυθούν από τα κράτη-μέλη ώστε να διορθωθούν, να βελτιωθούν τα συστήματα αυτό και ιδίω ομιλώ για τα πιο αυστηρά κριτήρια, τη μεγαλύτερη διαφάνεια των διαδικασιών, την αποφυγή των εκτονιστέρων τροποποιήσεων των συμβάσεων. Ε, πολλή δουλειά έχει γίνει σε όλες αυτές τις περιοχές. Και ήδη από το 2007 είχαμε καθορίσει μια τυπολογία παραβιάσεων και προτείναμε κατευθυντήριες γραμμές ε, επιδιόρθωσης. Αφενός προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι κίνδυνοι που μπορούμε να αποφύγουμε αλλά και αφετέρου προκειμένου να προταθούν οι απαραίτητες διορθωτικές δράσεις από τα κράτη-μέλη. Δουλεύουμε με τις αρχές, τις αρχές των κρατών μελών και σημείωσα ότι το ελεγκτικό συνέδριο πρώτο είχε εκδώσει ε, έκθεση ε, ελέγχου το 2004 υπό την έννοια αυτή εμείς συνεργαστήκαμε πολύ στενά με το συνέδριο για να έχουμε μια κοινή μεθοδολογία ιδιαίτερα στις δημόσιες συμβάσεις και από το 2011 έχουμε μοιραστεί με τις αρχές του ελεκτικού συνεδρίου το checklist που είχαμε σχετικά με τον έλεγχο που πρέπει να διεξάγεται και ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι ελεκτικές αρχές των κρατών μελών θα ακολουθούν αυτή την μεθοδολογία. Έχουμε αναπτύξει και οικοδομήσει μια εμπιστοσύνη αμοιβαία θα έλεγα επί τη βάση αυτών των κοινών αρχών και κανόνων και νομίζω ότι οι αρχές ελέγχου που είναι υπεύθυνε ε, ακολουθούν και ελέγχουν κατά τον τρόπο αυτό άνω του 90% των ε, πόρων των ταμείων. Εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε με τις υπόλοιπες για να βελτιώνουμε την μεθοδολογία και να εξασφαλίζουμε πάνω απ' όλα ότι χρησιμοποιούμε κοινή μεθοδολογία. Τώρα θα ε, ήθελα επίσης να τοποθετηθώ απέναντι σε κάποια μεγέθη, ευχαριστώντας και το συνέδριο. που δημοσίευσε στην ουσία μέσω της έκθεσής του το ελεγκτικό συνέδριο το σχέδιο δράσης μας γιατί στη σελίδα 43 περιγράφεται πάρα πολύ καθαρά το σχέδιο δράσης της Κομισιόν και δημοσιεύτηκε δηλαδή πριν το κάνουμε εμείς. Θα ήθελα όμως να επανέλθω σε κάποιες ιδέες που αναφέρονται εδώ όπως αυτό το 40% που αναφέρεται και αυτό είναι σαφές στην έκθεση πρόοδου, ιδιαίτερα στην ε, σελίδα 19 υπάρχει μια γραφική απεικονισή που ε, εξηγεί ότι αυτή είναι η συχνότητα των σφαλμάτων που παρατηρούνται ετησίως και ε, από το σύνολο αυτό των σφαλμάτων το 29% ήταν σοβαρά σφάλματα. Δηλαδή ο δικαιούχος δεν θα έπρεπε να έχει κερδίσει τον διαγωνισμό για παράδειγμα. Ή υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης στις υπόλοιπες περιπτώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος δημοσιονομικής διόρθωσης, ακόμα και αν υπάρχει κάποια έλλειψη συμμόρφωσης σε, κάποια, σε κάποιο στάδιο της ε, λυπής διαδικασίας. Σοβαρά σφέλματα θα είχαμε στην περίπτωση που έγινε ένα σφάλμα που δεν είναι αμεληταίο αλλά το οποίο δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα αν θέλετε της διαδικασίας του διαγωνισμού και της ανάθεσης. Στην ετήσια έκθεση λοιπόν του ετησίου συνεδρίου που παρουσιάστηκε στην, ε, στο Κοινοβούλιο την Τρίτη αναφέρει ένα συνολικό ποσοστό 4,4% και όχι σαν αυτά που ακούσαμε και παρουσιάζουμε εδώ και πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί με τη διάκριση αυτή. Επίσης ο κύριος Σόουεν ε, υποβάλλει και κάποια μεγέθη τα οποία διαβιβάζει από τα κράτη-μέλη, ε, τα οποία όμως κράτη-μέλη, 12.000 συνολικά παραβιάσεις, εκ των οποίων 2% αναφέρθηκαν ως υποψία παραβίασης και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δουν οι αρμόδιες αρχές κατά πόσο αυτό ισχύει. Δηλαδή πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τα μεγέθη που εμφανίζονται, αλλά δεν έχουμε πάντα να κάνουμε με απάτη. Υπάρχει ένα θέμα διαφθοράς στο σύνολο του ευρωπαϊκού εδάφους. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που μας δείχνουν ότι οι δημόσιες προμήθειες ιδιαιτέρως είναι συνδεδεμένες με υψηλό κίνδυνο διείσδυσης της διαφθοράς, αλλά περισσότερο έχουμε να κάνουμε με έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης, έλευση δυνατοτήτων σχετικά με τις ε, συνολικές ε, αναθέσεις και εργολαβίες από τοπικές αρχές που συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα να διοργανώσουν και να αναθέσουν όλα αυτά. Και υπάρχει λοιπόν ένας ενγενής παράγοντας κινδύνου. Πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε, να ταυτοποιήσουμε πολύ πιο προσεκτικά ή στις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη αυτό το δυναμικό, αυτή τη δυνατότητα που υπάρχει και να τους βοηθήσουμε να την βελτιώσουν. Και εμείς ελέγχουμε τους ευρωπαϊκούς ε, κανόνες, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους εθνικούς κανόνες. Εάν εκεί υπάρχει υπερβολική περιπλοκότητα που προστίθεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτό οδηγεί σε σφάλματα αυτό που λέμε gold plating δηλαδή στα ελληνικά. Ε, και εκεί υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης ώστε να μην είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως επί των θεμάτων αυτών. Γιατί και εδώ έχουμε ένα πεδίο πηγής πολλών σφαλμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο κύριος Νόνες Αλμέιδα Θέλω να πάρω το λόγο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο βασικός παράγοντας εδώ για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις είναι να υπάρξουν διοικητικές αλλαγές και αλλαγές σε ό,τι αφορά και την κουλτούρα που επικρατεί στη διοίκηση, να κατανοήσουμε ποιο είναι ο στόχος του συστήματος και των κανόνων για, την, ε, για τις δημόσιες συμβάσεις. Γι' αυτό λοιπόν συνεργαζόμαστε με τη Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο και ασφαλώς και με το Ελεκτικό Συνέδριο για να υπάρξει μια θεματική προσέγγιση με τα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν συστημικές δυσκολίες στις δημόσιες συμβάσεις. Και πιστεύουμε ότι καλό είναι να υπάρχουν και κυρώσεις, αλλά πολύ πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν και τα σωστά κίνητρα. Γιατί το βασικό είναι τα κράτη-μέλη να κατανοήσουν το όφελος ενός αποτελεσματικού συστήματος και μόνο τότε θα καταφέρουμε να περάσουμε τις αλλαγές. Άρα, τεχνική αρρωγή σε μεγάλο βαθμό, προληπτική δράση. Και υποστήριξη για ενέργειες επιτόπου. Και αυτά δεν είναι μόνο σχέδια, γίνονται στην πράξη μαζί με τη Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο βοηθούμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν το σύστημα δημόσιων συμβάσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα την περιπλοκότητα των κανόνων, η μεταρρύθμιση του 2014 περιλαμβάνει και μια προσέγγιση εργαλειοθήκης. Μεγαλύτερη ευελιξία, πιο πολλές δυνατότητες για τις αρχές ε, που παρέχουν τις συμβάσεις αλλά προαπαιτείται μεγάλη εκπαίδευση και κατανόηση σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να γίνουν καλά αντιληπτέ οι δυνατότητε. Κατά τρίτον, σε ό,τι αφορά τη σημασία των δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια στρατηγική λιπνενία αγορά προσφάτω, όπου και παρουσιάζονται ιδέες για τα δεδομένα και τι δημόσιε συμβάσει. Δίνουμε ένα αύσματα στα κράτη-μέλη να έχουν μετρό για συμβάσεις τέτοιες δημόσιες και για τις τροποποίησεις των συμβάσεων για την διαφάνεια και την διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων. Επίσης προωθούμε περισσότερες πληροφορίες για, τον, ε, για τους ελέγχους, ελέγχους και αυτοματοποιημένες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, τις εκθεωρήσεις, προκειμένου όλοι να γνωρίζουν τι αποτέλεσμα είχε ο έλεγχο Να προωθηθεί μια τέτοια κουλτούρα έλεγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτον, προωθούμε εργαλεία ανάλυσης και εντοπισμού ανομαλιών στο σύστημα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Και έτσι να δούμε ποια είναι τα συστημικά ευρεία θέματα και όχι τόσο ή σποραδικές, περιστασιακές παραβιάσεις. Άλλα δύο σχόλια για το διασυνοριακό εμπόριο και πώς, μάλλον τη διασυνοριακή διάσταση της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και τι κάνουμε για να την προωθήσουμε. Παρουσιάσαμε και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ ένα σύστημα το οποίο έχουμε αναπτύξει, το οποίο θα ευνοήσει και θα δώσει δυνατότητα σε μικρούς φορείς, όπως τους Ολλανδούς για παράδειγμα στο Βέλγιο, να συμμετάσχουν σε ένα δημόσιο διαγωνισμό με ένα ενιαίο έντυπο και όχι να αναγκάζονται να συμπληρώνουν πάρα πολλά έντυπα περίπλοκα. Για όλες λοιπόν τις διαδικασίες θα υπάρχει ένα ενιαίο έντυπο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν οι υποψήφοι προκειμένου να δούμε κατά πόσο πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια. Επίσης, ε, πράγματα τα οποία δεν εντοπίζονται συχνά, όπως η καλύτερη μετάφραση για τις ε, δημοσιεύσεις. Και εδώ γίνεται καλή δουλειά από την υπηρεσία δημοσίων συμβάσεων. Νομίζω ότι αυτό λοιπόν θα βελτιώσει πολύ καλύτερα τις δυνατότητες συμμετοχής σε όλη την Ευρώπη, σε τέτοιους διαγωνισμούς. Η Επιτροπός Μπρισχόσκα και η, η Γενική Διεύθυνση Γκρου είναι πολύ δραστήρια και σκοπεύουν να τα εφαρμόσουν όλα αυτά στην τρέχουσα θητεία με τη συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Ρίτζιο και με την υποστήριξη και αρρωγή ασφαλώς του Ελληνικού Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και όλους τους συμμετέχοντας στη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας, κύριε Όουν, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που μας επεξηγήσατε την έκθεση. Έχουμε συστάσει και το όραμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σχέδιο δράση το οποίο προτείνει. Βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογή. Και θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ελεκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή Ρέτζη θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαδικασία. Και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδατε άλλωστε και πόσο μας ενδιαφέρει το θέμα από τη συζήτηση που έγινε. Κατανοούμε λοιπόν την σοβαρότητα του θέματος και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να ξανασυναντηθούμε στο μέλλον με καλύτερα νέα, καλύτερε ειδήσει από τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Σα ευχαριστώ πολύ, λοιπόν, λέει η Πρόεδρο, και περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Ο δεύτερος ε, φιλοξενούμενός μας σήμερα το πρωί είναι ο κύριος Φρεντερίκ Βαλιέ, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, CEMR. Θα μας παρουσιάσει την τρέχουσα και τη μελλοντική δουλειά του Συμβουλίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1951. Είναι μια ε, ομπρέλα δημοκοινοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, έχει 60 μέλη και αντιπροσωπεύει 150.000 τοπικές ε, αρχές και φορείς. Στο site τους ε, λένε ότι έχουν διπλό ρόλο να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή πολιτική και η νομοθεσία σε όλους τους τομείς που έχουν άμεση επιπτώση σε δήμους και κοινότητες και δεύτερον να αποτελέσει ένα φόρουμ συζήτησης και διαλόγου μεταξύ των ε, τοπικών και περιφερειακών αρχών με τους εθνικούς ε, φορείς σε κάθε περίπτωση. Η CMR μας επισκέφθηκε για τελευταία φορά το 2011 Λυπάμαι πολύ που πέρασε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να τους ξαναφιλοξενήσουμε. Είναι ευκαιρία λοιπόν τα νέα μέλη της ε, Επιτροπής ε, Περιφέρειας Ανάπτυξης να μιλήσουν, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους αυτούς που εκπροσωπούν τόσους τοπικούς φορείς. Έχουμε περίπου μία ώρα στη διάθεσή μας. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στην, καταρχήν στον κύριο Βαλιέ για να μας παρουσιάσει περίπου για 15 λεπτά, αν σας αρκεί κύριε Βαλιέ, αυτό το χρονικό διάστημα ε, τις ε, δραστηριότητες του CMR και μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να παρουσιάσω το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης ε, εδώ στα μέλη της Επιτροπής. Είναι ε, το, η πιο πλατιά και η πιο παλιά ευρωπαϊκή οντότητα που αντιπροσωπεύει δήμους και ε, περιφέρειες. Ε, αντιπροσωπεύουμε χώρες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σίγουρα όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 41 συγκεκριμένα χώρες έχουν μέλη ε, στο CMR. Ε, θέλουμε να προωθήσουμε μια ενιαία ειρηνική και δημοκρατική Ευρώπη θα βασίζεται στις τοπικές κυβερνήσεις, σεβόμενες αρχές επικορικότητας και την συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το CMR είναι αναγνωρισμένος ως κοινωνικός εταίρος στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο, αντιπροσωπεύοντας τοπικές ε, κυβερνήσεις ε, ε, ως εργοδότες. Αυτό επιβεβαιώθηκε από την έκθεση της Eurofound που έγινε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Είμαστε μόνιμοι ε, παρατηρητές στο Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς επίσης και σε πολλά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι που είμαι εδώ για να ανταλλάξουμε απόψεις με την Επιτροπή. Όπως είπατε και εσείς, τελευταία φορά που ήμασταν εδώ ήταν το 2011. Παρόλο που είμαστε σε τακτική επαφή με πολλά από τα μέλη της Επιτροπής σας, ε, με, ο κ. Σάλμπρεκτ για παράδειγμα, ήταν αντιπρόεδρος της, ε, του CMR πριν γίνει ευρωβουλευτής. Ε, είμαστε φίλοι, ο κ. Φανίστελ Ρόι επίσης, η κ. Μπρέσελ ε, και πολλοί άλλοι, πολλά άλλα από τα μέλη σας είναι άνθρωποι με τους οποίους είμαστε σε στενή επαφή και μερικές φορές και φίλοι. το CMR είναι και το ευρωπαϊκό κλιμάκιο του Παγκόσμιου Διοργανισμού πόλεων και τοπικών κυβερνήσεων το οποίο μας εκπροσωπεί σε διεθνές επίπεδο στον Οργανισμό Εθνών και αλλού. Σε, για παράδειγμα, ε, διοργανώνει, ε, ε, μας, συγγνώμη, μας αντιπροσωπεύει, θα μας αντιπροσωπεύσει στην ΚΟΠ, στην, στο Habitat 3 και του χρόνου κλπ ε, καλύπτουμε ένα ευρύ πεδίο από την διακυβέρνηση, τη δημοκρατία και ε, την ε, ηθαγένεια. Ε, είμαστε μία από τους πιο βασικούς φορείς που προωθούν την συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ε, μετά, εδώ και αρκετά χρόνια εφεύραμε και αναζωογονήσαμε ε, το θεσμό της αδελφοποίησης. Ε, επίσης ε, την χάρτα ε, ποιότητας της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ε, η οποία έχει υπογραφεί από 1500 ε, τοπικές οργανώσεις και φορείς στην Ευρώπη. Είμαστε το, στην πρώτη φάση της σύνταξης και υιοθέτησης της ε, χάρτας των τοπικών κυβερνήσεων στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ε, το 1953 ήδη είχαμε υιοθετήσει το χάρτη των τοπικών ελευθεριών. Ένα άλλο κλάδο δράση, τομέα δράση, είναι η διαχείριση των δημοσίων υπηρεσιών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και η σχέση με τον κοινωνικό διάλογο και την διαχείριση των δημοσίων πολίων σε τοπικό επίπεδο. Ένα άλλο ζήτημα είναι η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και η περιφερειακή ανάπτυξη. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε και επιθυμούμε διακόπω να συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή σας στην ανάπτυξη και την προώθηση νέων ιδεών για το πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ε, τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και ταυτόχρονα ε, να χρησιμοποιηθούν σωστά. Οι δημογραφικές ε, αλλαγές που παρατηρούν σε αυτό το τομέα είναι κάτι που παρακολουθούμε πολύ στενά. Το περιβάλλον, το κλίμα και η ενέργεια είναι άλλο κεφάλαιο των δραστηριοτήτων μας. Σας ανέφερα την ΚΑΠ 21 προηγουμένως, στην οποία συμμετέχουμε. Συμμετέχουμε επίσης και στην, στο Σύμφωνο των Δημάρχων ε, για την ε, μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και την αύξηση των, της χρήσης των ανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ε, είμαστε τμήμα του Consortium που διοργανώνει την σύνοδο των δημάρχων και εμπλεκόμαστε και σε άλλα project σχετικά σχετικά με την, προς, με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το City Invest για παράδειγμα που επενδύει στην, σε ανώσιμες πηγές ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, τέλος, είμαστε το ευρωπαϊκό, ο ευρωπαϊκός κλάδος του, UCLG που είναι το παγκόσμιο, η παγκόσμια ομπρέλα δήμων και περιφερειών το Συμβούλιο είναι, ε, αποτελεί πλατφόρμα κεντρική συνεργασία Δήμων και Περιφερειών ε, που προωθήθηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει την αποκεντρωμένη συνεργασία μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων και το, των αντίστοιχων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, το, στην αρχή 2015 α, υπογράψαμε μια στρατηγική εταιρική σχέση με την Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ, ε, Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Ορισμένα επίγοντα ε, και επίκαιρα θέματα που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Πρώτον, η, κρίση, η μεταναστευτική κρίση, ε, ε, η προσφυγική κρίση για την ακρίβεια. Ενημερώσαμε ήδη από την περασμένη άνοιξη την Κομισιόν για τις ε, συνέπειες κατάσταση που μπορεί να έχει κατάσταση στη Μεσόγειο επί των τοπικών κυβερνήσεων. Είμαι σίγουρος ότι όλοι γνωρίζετε πως οι πρώτοι εμπλεκόμενοι στο, στο θέμα του προσφυγικού είναι οι δήμοι και οι κοινότητες στη Μεσόγειο, αλλά προφανώς όχι πια μόνο στη Μεσόγειο, παντού σε όλη την Ευρώπη. Ε, Ε, συνεργαζόμαστε με τα μέλη μας έτσι ώστε να αξιολογήσουμε και να αναλύσουμε την κατάσταση. Έχουμε κάνει μάλιστα και μια έρευνα. Ε, αν μπείτε στο site μας μπορείτε να τη βρείτε αν ενδιαφέρεστε. Και συζητούμε με τη Γενική Διεύθυνση Home Εσωτερικών Υποθέσεων για να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις, ε, ε, τους Δήμους και τις κοινότητες, την τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, πιέζουμε έτσι ώστε ε, χρηματοδότηση να δοθεί στους Δήμους και τις κοινότητες, ίσως όχι κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, γιατί οι κανόνες δεν το ε, επιτρέπουν, αλλά τουλάχιστον να δοθεί στα κράτη-μέλη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται σε τοπικό επίπεδο από, το, από τις ροές. Έχουμε συμμετάσχει δραστήρια τα δύο τελευταία χρόνια όπου συζητούμε τιντούνται θέματα συνοχής και διαφορετικών ταμείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε ότι θα συνεργαστούμε με τον Γιάννο Όλμπρεχτ στην διάμεση, στη σύνταξη της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης. Θέλουμε να να ε, θίξουμε τέσσερα βασικά ζητήματα σε σχέση με αυτό. Θέλουμε να ενισχυθεί η αρχή της ε, συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης που ήδη βρίσκεται στο πρόγραμμα. Θέλουμε να δοθεί μεγαλύτερη σημασία σε αυτό. Να στηριχθεί η τοπική ανάπτυξη. Επιμένουμε για αυτό το θέμα εδώ και πολλά χρόνια και στηρίζουμε ασφαλώς και τα ε, ολοκληρωμένα εργαλεία, ε, εδαφικά εργαλεία. Σε ό,τι αφορά τα επιχειρησιακά προγράμματα ε, έχουμε ε, συντάξει διάφορες εκθέσεις και μελέτες. Οι δύο πιο πρόσφατες είναι η επισκόπηση της εφαρμογής των τοπικών σχεδίων επενδύσεων από τα κράτη-μέλη και η ανάλυση της συμμόρφωσης με τις αρχές ε, εταιρική σχέση των ε, προγραμμάτων συνοχής ε, και ε, περιφερειακής ανάπτυξης. Έχω αντίγραφα, αν θέλετε μπορώ να σας δώσω. το CMR είναι μια από, ένας από τις φορείες που συμμετέχουν στο φόρουμ για την αστική ανάπτυξη συμμετέχουμε και στις άτυπες συνεδρίες των ε, Συμβουλίων Υπουργών, των διαφόρων Προεδριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεισφέρουμε στην ε, μελλοντική ε, αστική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα με τη στήριξη των Ολλανδών Υπουργών, του Ολλανδού Υπουργού, γιατί, που, στη σύνταξη ενός κειμένου που θα επηρεάσει ελπίζω την Ολλανδική Προεδρία. Η ανακοίνωση των Υπουργών της ε, Ρίγα, των Υπουργών στη Ρήγα ε, τον περασμένο Ιούνιο αναγνώρισε το CMR στο ρόλο του η δική μας ε, προσέγγιση είναι πολύ συγκεκριμένη σε ό,τι αφορά την εδαφική και τοπική συνοχή λίγο διαφορετική από αυτήν της Eurocities. Καλωσορίζουμε την ε, προσέγγιση που ε, λαμβάνει υπόψη και την ε, συμπληρωματικότητα μεταξύ αστικών και μυαστικών περιοχών. Συνεισφέρουμε επίσης στον διάλογο για την απλοποίηση και τη μείωση της γραφειοκρατίας στα ευρωπαϊκά ταμεία. Είμαστε ε, μία, ένας από τις τέσσερις φορείς που κλήθηκαν να υποβάλουν τις, να παρουσιάσουν τις απόψεις τους ε, στις 15 Οκτωβρίου από την, ε, στην ακρόαση της Επιτροπής Ρέτζι. Ε, έχω αντίγραφα της παρουσίασής μας για όσους ενδιαφέρονται. Σύντομα θα ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε την μελλοντική πολιτική συνοχή για τα έτη μετά το 2020. ετοιμάζουμε ε, το επόμενο συνεδρίο μας τον Απρίλιο και ήδη έχουμε ξεκινήσει ένα διάλογο, ε, μια διαβούλευση. Ε, ζητούμε τις απόψεις τοπικών και περιφερειακών ηγετών, αλλά η διαβούλευση να ανοιχτεί και στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε να δούμε ποιο θα είναι το όραμά μας για την τοπική και περιφερειακή οργάνωση και κατάσταση για την περίοδο μέχρι το 2030. θα ε, προκύψει μια έκθεση την οποία θα, ανα... αποστείλουμε στην συζήτηση για την Ευρώπη του 2030 κάποια στιγμή την Άνοιξη. Το CMR ε, είναι προσιλωμένο στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη και σε συνεργασία με, την με τη γαλλική κυβέρνηση ε, εργαζόμαστε επί μιας πιο φιλικής ε, ε, εκδοχής ε, του εγχειριδίου για την, ανάπτυξη των, την αστική ανάπτυξη. Θα στηθεί το 2016 στην Λευκοσία. Θα αφορά κυρίως μικρές και μεσαίες πόλεις για να τις βοηθήσει να ακολουθήσουν μια βιώσιμη ανάπτυξη. Το CMR ως Ευρωπαϊκό Κλιμάκι του UCLG εμπλέκεται σε συζητήσεις και σε διεθνές επίπεδο ε, στον ΟΗΕ, είμαστε μέλη της Παγκόσμιας Task Force για την τοπική περιφερειακή κυβέρνηση, συμμετέχουμε στην ε, προετοιμασία της ε, αντισιακής ατζέντα του ΟΗΕ για μετά το 2015, στους βιώσιμους αντισιακούς στόχους και στην δημιουργία μιας καινούριας αστικής ατζέντα στον ΟΗΕ που θα συμφωνηθεί στο Habitat 3 το 2016 στο Ιμπογκοτά. Η συνάντηση προετοιμασία θα λάβει χώρα στην Πράγα το Μάρτιο και ασφαλώς θα είμαστε και εμείς εκεί. Τα περιεχόμενα αυτών των ε, θεματικών ενωτήτων ε, το Τοπικές και προσωπικές κυβερνήσεις ε, συνεργάζονται μέσω αυτών ε, μεταξύ τους ε, και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρόθεση είναι η ευρωπαϊκή ατζέντα ε, να ενταχθεί στην παγκόσμια ατζέντα και θα εστιάσουμε σε δύο από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης κυρίως. Ε, οι βιώσιμες ε, κοινότητες και πόλεις είναι ο στόχος 11 που είναι προφανώς ο πιο κέριος στόχος για μας, ο πιο σχετικός και τον στόχο για την διακυβέρνηση που είναι ο υπαριθμό 16 έτσι ώστε οι συμφωνίες που ε, συνάπτονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, θα συνάδουν με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ε, το CMR ενδιαφέρεται, επίσης, ενδιαφέρεται προφανώς για μια επικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και το διακομματικό, διακομματική ομάδα Urban και ελπίζουμε ότι θα βρούμε έναν τρόπο να ε, ενημερώνετε η Επιτροπή σας άμεσα για τις θέσεις μας. Θα θέλαμε επίσης να καλέσουμε τα μέλη της Επιτροπής σας που ενδιαφέρονται να έρθουν στο συνέδριο μας στη Λευκοσία τον Απρίλιο του 2016. Αυτό το συνέδριο είναι η βασική, το η κύρια συνάντηση μεταξύ τοπικών ηγετών. Περίπου χίλιοι δήμαρχοι, και γενικότερα πολιτικοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη θα έρθουν εκεί, υπολογίζουμε, περιμένουμε και εσάς, προφανώς μέλη του Κοινοβουλίου και μέλη της Επιτροπής, καθώς επίσης και ηγέτες από όλη την Ευρώπη. Ο βασικός μας ε, στόχος, όπως είπα προηγουμένως, είναι η Ευρώπη 2030. Θέλουμε να χτίσουμε ένα όραμα η Ευρώπη των τοπικών και περιφερειακών αρχών με περισσότερη αισιοδοξία πλέον. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε για τις προσκλήσεις. Προφανώς έχετε συμμετέχοντες ε, και εκπροσώπους στην Επιτροπή μας ε, που ασκούν επιρροή και lobbying. Ε, Συνάδελφοι, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, ο κύριος Όλμπριχ. Ναι, εκ μέρους ε, του λόμπινγκ ακριβώς ε, της CMR και ως πρώην αντιπρόεδρος να θυμίσω ότι υπήρξε πολύ δραστήρια η CMR σε ένα από τα προγράμματα και προετοιμάζοντας και την όλη έννοια και ιδέα της Επιτροπής των Περιφερειών. Το σχόλιο μου προς το Γενικό Γραμματέα είναι το εξής. Θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή παλιά η συζήτηση ήταν κατά πόσον οι διάφορες εθελοντικές οργανώσεις όπως η CMR που είχε ξεκινήσει το 50 με το συνέδριο των ε, δημάρχων που ήθελαν να εκπροσωπήσουν την, ε, το σύνολο τέλο πάντων της Ευρώπης χρειαζόμαστε, είναι η ερώτησή μου, τους διάφορους αυτούς θεσμούς, φορείς, ενώσεις, εφόσον έχουμε την Επιτροπή των Περιφερειών. Γιατί εφόσον η Επιτροπή των Περιφερειών εκφράζει όλες τις τοπικές λογικότητες, τι εκφράζουν αυτές οι ενώσεις. Η εμπειρία λοιπόν μας δείχνει ότι υπάρχουν διαφορετικές εμπειρίες και χρειαζόμαστε και τις δύο, και τα δύο επίπεδα εκπροσώπησης. Εσείς όμως Γενική Γραμματέα πώς βλέπετε την διάκριση της εκπροσώπησης μεταξύ των δύο ή το συσχετισμό. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει επικάλυψη στην πραγματική εκπροσώπηση. Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η εκλεγμενη αντιπρόσωποι των τοπικών εκπροσώπων. Οι ενώσει είναι εθελοντικές οργανώσεις που εκπροσωπούν και μη κράτη-μέλη. Αλλά είναι πολύ σημαντικά, σημαντική αυτή η διάθρωση, ιδιαίτερα στο διάλογο με τα θεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή λοιπόν ήταν η ερώτηση, η σχόλιο μου. Ευχαριστούμε η κυρία Μαλέτιτς. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίζω τον Γενικό Γραμματέα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις θεματικές τις οποίες αναφέρθηκε εγώ ήθελα να αναφερθώ λίγο στην ε, μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη είναι οργανωμένα με διαφορετικό τρόπο εσωτερικά και πολλές, σε πολλά μάλλον από τα κράτη-μέλη οι περιφέρειες είναι μια πολύ σημαντική διάσταση για την υλοποίηση των ε, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, των επενδύσεων, τίποτα δεν μπορούμε να επιτύχουμε χωρίς την ισχυρή και ενεργό συμμετοχή των περιφερειών. Και έχω την αίσθηση ότι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς σκεφτόμαστε ακόμα αρκετά κεντρικό παγός αν θα έλεγα, αν θα μπορούσα να το πω έτσι. Σας ευχαριστώ κυρία Μαλετίτσου, έχουμε άλλες ερωτήσεις. Κύριε Ζούς, ε, ε, μία ερώτηση που έχει σχέση με τις ανησυχίες του CMR για την βιώσιμη ανάπτυξη. Πέρσι, το Σεπτέμβρη, κάποιες χώρες καθόρισαν 17 στόχους στους οποίους δεσμεύτηκαν για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Το CMR γνωρίζουμε ότι έχει εργαστεί επί μακρόν για τέτοιου είδου θέματα μέσω ε, εκδηλώσεων που έχει οργανώσει κλπ. Η ερώτηση είναι τι προτείνει το CMR σε ό,τι αφορά την σύγκρουση και την αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στις επιθυμίες, τα λόγια και, στην, και στις πράξεις. Ιδιαίτερα για χώρες οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, πώς μπορούμε να περάσουμε τις επιθυμίες στην πράξη. Ευχαριστώ. Thank you. The next question Ευχαριστώ. Ο κύριος Πολτσακ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτή που είχαμε του γραμματέα του Συμβουλίου. Εγώ ήμουν πρόεδρος της δεύτερης μεγαλύτερης ένωσης στην Τσεχία που εκπροσωπεί τους Δήμους. Και τώρα διερωτόμαστε πώς οι πόλεις, οι δήμοι θα έπρεπε να προετοιμαστούν για τον αντίκτυπο, τον όλο και αυξανόμενο της προσφυγικής κρίσεως. Μας δώσατε κάποια παραδείγματα, αλλά θα ήταν πολύ χρήσιμο να ακούσουμε και άλλα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάνσκουρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του CMR για την πλήρεστατη αυτή παρουσίαση και για την ενημέρωση που μας έκανε σχετικά με τις δραστηριότητες ε, του φορέα αυτού με τους Δήμους και τις περιφερειές για τις απομακρυσμένες ε, περιφέρειες πώς ενεργείτε ώστε να είστε σε συνεχή επαφή και να τις λαμβάνετε υπόψη στη δουλειά σας και τη δραστηριότητά σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βανίχτερόι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την δυνατότητα που μας δίνετε να βάλουμε το θέμα αυτό στην ατζέντα μας. Η οργανώσεις ε, οι οποίες διοργανώνουν ε, τέτοιες δράσεις ε, και που εκφράζουν την άποψη των πολιτών. Μία ερώτηση έχω να κάνω σε ό,τι αφορά το σύμφωνο του Άμστερνταμ. Προσφάτως, στις ημέρες ανοιχτών θηρών, στην συνεδρίαση με την Επιτροπή Περιφερειών, συμφωνήσαμε για ένα επί ενός οδικού χάρτη που θα κινείται προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της συζήτηση για την οριζόντια αστική ατζέντα. Και αυτά έχουν ενσωματωθεί σε ένα σύμφωνο του Άμστερνταμ, όπως ονομάζεται. Μία επεξήγηση των αποφάσεων του Συμβουλίου που περιλαμβάνει και μία δέσμευση των οργανώσεων που τοποθετούνται στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Αυτό ισχύει και για την δική σας οργάνωση. Η δέσμευσή σας στο δικό σας έργο πιστεύετε ότι επηρεάζει την ποιότητα της αστικής ατζέντα. Πρόκειται για ένα εργαλείο, ένα μέσο το οποίο προωθήσαμε εμείς το σύμφωνο λοιπόν του Άμστερνταμ. Ποια είναι η αποψή σας. Σα ευχαριστώ. Λέει Πρόεδρος, παρατήσεις. Ο κύριος Βαλιά λοιπόν έχει και πάλι το λόγο για να απαντήσει και να σχολιάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Για την πρώτη ερώτηση του Γιάνν Ολμπρέχτ για τη συμπληρωματικότητα μεταξύ ΚΟ και ΣΥΜΑΡ. Αυτό υπήρχε ω σχέση στην αρχή, αλλά με την πάροδο του χρόνου και των ετών θεωρώ ότι βρέθηκε μια καλή συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, των δύο οργανώσεων. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελεί μια συνέλευση, αν και δεν είναι εκνευριστική συνέλευση όπω το Κοινοβούλιο. Είναι μια συνέλευση λοιπόν που παρέχει απόψει ε, για του κανονισμού οι οποίοι ήδη βρίσκονται στη φάση τη εφαρμογή ενώ το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών είναι μια οργάνωση που λογικά δραστηριοποιείται σε πρώτερο χρονικό σημείο και δουλειά μας είναι να ακουστεί η φωνή της περιφέρειας στη φάση της κατάρτισης της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και γι' αυτό λοιπόν συνεργαζόμαστε σε πρώιμη φάση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με το Ευρωπαϊκό Κοινόβουλιο προκειμένου να ακουστούν οι απόψεις μας και να συνεργαστούμε για την καλύτερη δυνατή συνεργασία για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι η βασική διαφορά, θεωρώ εγώ. Φυσικά συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την Επιτροπή των Περιφερειών για μια μεγάλη σειρά θεμάτων και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να διευκρινίσουμε αυτό το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ μας. Κατά τη γνώμη μου όμως δεν υπάρχει οποιοδήποτε ανταγωνισμό μεταξύ των δύο σωμάτων. Μία καλή συμπληρωματικότητα μόνο θα πρέπει να εξευρεθεί. Και αυτό ισχύει και με άλλους οργανώσεις. Φυσικά είμαστε η μεγαλύτερη οργάνωση και τα μέλη μας ε, είναι στις εθνικές ενώσεις. Είναι λίγο διαφορετικά λοιπόν τα πράγματα σε σχέση με άλλες οργανώσεις που πραγματεύονται συγκεκριμένα θέματα. Αλλά ο ρόλος του CMR θεωρώ ότι είναι πιο πολύ σαν μια οργάνωση ομοσπονδίας. Έχουμε τη δυνατότητα να συνενώσουμε όλους τους φορείς την τράπεζα των διαπραγματεύσεων για να βρούμε τον κοινό τόπο. Και αυτό ισχύει όλος ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά την κρίση των προσφύγων στην παρούσα φάση, όπου μπορούμε να βάλουμε όλους τους ε, παράγοντες την ίδια αίθουσα για να βρούμε τις κοινέ τοποθετήσεις. Και αυτό με φέρνει στο θέμα τη σχέση του Συμβουλίου με το περιφερειακό επίπεδο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώνουμε ότι η σχέση επικεντρώνεται υπερβολικά πολύ στο κεντρικό επίπεδο το, από το ευρωπαϊκό επίπεδο στο κράτος μέλος. Και αυτό ασφαλώς προσπαθούμε να το αλλάξουμε, να το αντιμετωπίσουμε στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τοπικών και περιφερειακών και αυτοδιοικήσεων. Εμείς πιστεύουμε, και αυτό το αναφέρουμε παντού, ότι η μελλοντική ανάπτυξη, εξέλιξη της Ευρώπης αλλά και των άλλων επίρων εξαρτάται από την ικανότητα των περιφερειών και των ε, τοπικών αυτοδιοικήσεων να δημιουργήσουν δυναμικό ανάπτυξη. Και χρειάζεται η συμμετοχή των Δήμων και κοινοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κανονισμοί πολύ συχνά διοχετεύονται προς τις κεντρικές κυβερνήσεις και όχι προς τις περιφέρειες, προς τους δήμους, τις κοινότητες. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει ασφαλώς τα επόμενα χρόνια. Να συμπεριληφθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση στη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αναφέρθηκε, και στις συνθήκες ότι οι τοπικές κυβερνήσεις και οι περιφέρειες αναγνωρίζονται ως τμήμα της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης, αλλά θα πρέπει να αποκτήσει σάρκα και ώστα πλέον. Αυτό λοιπόν το στέλνουμε ως μήνυμα κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι τόσο προς το Κοινοβούλιο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας. Τώρα οι στόχοι της ε, βιώσιμης ανάπτυξης ε, στις ε, οποίες αναφερθήκατε κύριε Ρουάσκ, Δουλέψαμε πολύ επί των στόχων αυτών, αναφέρθηκα στον 11 και τον 16, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι, εντός των οποίων καλούνται οι τοπικές ε, αρχές να έχουν συγκεκριμένη δράση και δραστηριότητα. Και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταλάβει ότι προκειμένου να επιτευχθούν διάφοροι ευρείας κλίμακα στόχοι πρέπει να κινητοποιηθούν οι τοπικές αρχές. Το 100% του παγκόσμιου πληθυσμού θα, μένει σε, θα ζει σε πόλεις ε, όπως δείχνουν οι προβολές και οι εκτιμήσεις σύντομα. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα συμπληρωματικότητος μεταξύ των αστικών περιοχών και των περιοχών της υπαίθρου. Έχουμε ένα πρότυπο δημοκρατικής διακυβέρνησης που μπορούμε να διαβιβάσουμε στον κόσμο χωρίς να θέλουμε να δίνουμε μαθήματα σε κανέναν αλλά έχουμε κάποιες δομές ε, δημοκρατικής εκπροσώπησης και διαλόγου που θα πρέπει να κατευθύνουν τη δράση μας παγκοσμίω. Βεβαίως μεταξύ των προθέσεων και της πράξης ε, υπάρχει απόσταση. Οι στόχοι της χιλιετίας δεν έχουν επιτευχθεί για παράδειγμα ε, ή η στρατηγική του 2020 δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε τους στόχους αυτούς. Αλλά πρέπει να θέτουμε συνεχώς μακροπρόθεσμους στόχους προκειμένου τουλάχιστον ένα τμήμα αυτών να το πετυχαίνουμε. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση είναι προφανώς ε, ένα τεράστιο ζήτημα, ένα τεράστιο διακύβευμα. Εμείς ε, στο πλαίσιο αυτό έχουμε κάνει πάρα πολλές αναρρυθμίτες ε, μελέτες, ιδιαίτερα η τελευταία του 11 2012 ήταν ε, σχετικά με τις δημοσιονομικές δραστηριότητες των τοπικών φορέων και αυτό το παρακολουθούμε ζωηρά. Και έχουμε και προτάσεις για την καταπολέμηση της κρίσεως ακριβώς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επ' αυτού συνεργαστήκαμε με τους ε, Πορτογάλους, Έλληνες, Ιταλούς ε, και Ισπανούς ε, συναδέλφους για να το αναπτύξουμε αυτό το ζήτημα σε εθνικό επίπεδο. Για την προσφυγική κρίση αναφέρθηκα βεβαίως. Είχαμε κάνει μια πρώτη έρευνα σχετικά με την κατάσταση των δημοτικών και περιφερειακών κυβερνήσεων. Αυτό έχει διαχυθεί και στην τσεχική δημοκρατία και σε άλλες ε, κεντροευρωπαϊκές χώρες είναι πλέον κρίσιμη η κατάσταση. Αυτό που θα θέλαμε να προτείνουμε και προτείναμε ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν η ανάπτυξη κάποιων καθητηρίων γραμμών πώς μπορούν να φιλοξενούνται οι πρόσφυγες τοπικά καλύτερα και θα θέλαμε να αναπτύξουμε και να φιλοξενήσουμε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής βελτίστων πρακτικών σε αυτό γιατί σε πολλές χώρες στα νεότερα δηλαδή κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τοπικές κυβερνήσεις δεν έχουν τέτοια εμπειρία φιλοξενίας και εγκατάστασης τέτοιων αριθμών προσφύγων και μεταναστών. Υπάρχουν λοιπόν εντάσεις, υπάρχουν θέματα που θα πρέπει να τα καλύψουμε, αυτό θα το κάνουμε στους ερχόμενους μήνες, αλλά θα θέλαμε να επιμείνουμε ότι οι πόλεις και οι τοπικές κυβερνήσεις πρέπει να έχουν το χρόνο και τα μέσα γιατί έχουν τη βούληση αλλά πρέπει να έχουν και τα μέσα να φιλοξενήσουν τους αριθμούς των ανθρώπων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν και οι κεντρικές εθνικές κυβερνήσεις να αναλάβουν το ρόλο που τους αντιστοιχεί. Το θέμα των ε, από μακρισμένων περιφερειών να πω στον αγαπητό εκπρόσωπο είναι κάτι που βεβαίως καθότι είστε γαλλόφωνος και σας το λέω γαλλικά έχουμε μια ένωση γαλλοφώνων περιφερειών της Ευρώπης η οποία παρεμβαίνει τακτικά στα υπερπόντια εδάφη και περιφέρειες για να υποστηρίξει τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στην χρηματοδότηση ίσως θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα. Αλλά υπάρχει ε, ένωση που εκπροσωπεί ακριβώς τις ε, υπερπόντιες περιφέρειες, ε, ίσως θα έπρεπε να κάνουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Επ' αυτού με μεγάλη χαρά θα συμφωνούσα να αναλάβουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Και για την τελευταία ερώτηση του κυρίου Βανίστελ Ρόι. Ελπίζουμε ότι η επόμενη, το επόμενο αστικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναφέρεται στην σχέση των ευρωπαϊκών θεσμών και πόλεων και δήμων. Βέβαια δεν είναι σαφές πώς αυτό θα οργανωθεί. Δεν είναι σαφές πόσα κράτη-μέλη θα υποστηρίξουν το αστικό θεματολόγιο. Υπάρχει ακόμα αντίσταση, όπως θα γνωρίζετε. Το προσπαθούμε και από κοινού με τους υποστηρικτές της πρωτοβουλίας αυτής ε, ελπίζω και πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε μια καλή πρόταση και βεβαίως σε συνεργασία με τα Ολλανδικά, Γαλλικά και Γερμανικά αρμόδια Υπουργεία και φορείς αλλά η μελλοντική αστική ατζέντα, το αστικό θεματολόγιο δεν θα πρέπει να τεθεί σε ανταγωνισμό προς την περιφερειακή πολιτική σε καμία περίπτωση. Πρέπει να την συμπληρώνει ακριβώς στο επίπεδο της, ε, του συσχετισμού της δομής μεταξύ των περιφερειών και των πόλεων. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε και στην CMR να επιτύχουμε. Ευχαριστώ λοιπόν Πρόεδρε και βεβαίως είμαι στη διάθεση όλων των μελών σας οι υπηρεσίες μας ε, είναι εδώ στις Βρυξέλλες για να υπηρετούν και εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ ίδια. Ελπίζω ότι θα παραμείνουμε σε στενή συνεργασία στο μέλλον και θα μας ενημερώνετε για τις επιτυχίες σας και για το πώς εκπροσωπείτε τις ε, τοπικές αρχές ε, πώς είστε η φωνή τους. Θα είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Ας περάσουμε το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Είχαμε προγραμματίσει τις για τις 11 και 4. Έχουμε λοιπόν μερικά λεπτά ακόμα. Να περιμένουμε και τα υπόλοιπα μέλη, τρία λεπτάκια. Ωραία. Αν χρειάζεται τρία λεπτά, θα ε, διακόψουμε και θα μιλήσουμε μεταξύ μας. Προετοιμάστε μεταξύ και την κάρτα ψηφοφορία σας. Okay, colleagues. 11.15. Ωραία. Κάντε και τέταρτο. Ξεκινάμε τις προφορίες. Ξεκινώντας με την Ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την έκθεση του 2014 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Από το 2013 η ΚΟΝΤ και η ΕΚΟΝ ε, συντάσσουν γνωμοδότηση ε, πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ε, Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών είναι υπεύθυνη. Ο στόχος της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Με τη νέα γενιά της, ε, των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης ε, που χρειάζονται, έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σηματοδότησης. Ο κύριος Γιάκοψιτς είναι ο εισηγητής μας. Μέχρι την προθεσμία της 21ης ε, Οκτωβρίου 53 τροπολογίες είχαν υποβληθεί ενώ ο εισηγητής υποβάλλει μερικές δικές του τροπολογίες συμβιβασμού. Κύριε Γιάκοψιτς, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλες που συνεργάστηκαν μαζί μου παρόλο ότι επικράτησαν και κάποιες εντάσεις, μικροεντάσεις, πιστεύω ότι η έκθεση είναι τελικά καλή, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλα τα στοιχεία όλοι μας, όμως η έκθεση αυτή βλέπει λίγο διαφορετικά με έναν πιο καινοτόμο τρόπο το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ζητούμε ένα καινούριο ρόλο για αυτήν, ένα ρόλο που θα ε, Ε, βοηθά τους ε, ε, οικονομικού οικονομικούς φορείς αλλά και τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ωραία. Ας περάσουμε στην ψηφοφορία. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ετήσια έκθεση 2014. Τροπολογία υπαρθμών 1. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τροπολο, ε, τροπολογία, συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Υπαριθμόν τρία συμβαστική τροπολογία υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Χωριστή ψηφοφορία. Το την οποία ζήτησαν οι φιλεύθεροι. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 29 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Για αλλάξτε θέση. Ε, δουλεύει εκεί. Περνάμε στην τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Και πάλι ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Τροπολογία 31. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία, συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. απόχέ. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, Σημαντική τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Η νομοδότηση εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Γιάκοψιτς. Και τώρα συνεχίζουμε με την δεύτερη έκθεση, την δεύτερη ψηφοφορία. για την γνωμοδότηση για την ετήσια έκθεση του 2014 για την ε, προσπάθεια των οικονομικών συμφερόντων κατά πολέμηση της απάτης. Τον Ιούλιο η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων συμπεριλαμβανομένης και της καταπολέμησης της απάτης. Η Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού είναι η Καθελήνα Αρμόδια, η Ρέτζη Γνωμοδοτή. Στις 15 Οκτωβρίου ο κύριος Βόνο, ο εισηγητής μας, παρουσίασε την, το σχέδιο έκθεσης, το σχέδιο γνωμοδότησης και έχουν ε, κατατεθεί 51 τροπολογίες. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Βόν θα ήθελε να πάρει το λόγο, να πει δύο λόγια πριν ξεκινήσουμε την, τροπο, την ε, ψηφοφορία. Εν συντομία, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τους κύριους εισηγητές για την, για την βοήθειά τους, την υποστήριξή τους θα δούμε οι συνάδελφοι ότι πιο πολλές ε, τροπολογίες έχουν ενσωματωθεί σε 10 συμβιβαστικές τροπολογίες και αυτό καταδεικνύει το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των ομάδων και κατά πόσο συγκλίνουν οι απόψεις στην Επιτροπή και σε ό,τι αφορά θέματα καταπολέμησης απάτης. Όλοι θέλουμε να διασπαλίσουμε ότι τα χρήματα και τα κονδύλια τα πάνε με τον τρόπο. Αυτά λοιπόν αποτυπώνονται στι 10 συμβαστικέ τροπολογίε. Μάλιστα λοιπόν, λέει ο πρόεδρο, να ψηφίσουμε. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Απόχε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική 8, τροπολογία 8 μάλλον υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, Αποχέ. απορρίπτεται. Συμβαστική 4, υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβασμό 5, υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Θα χρειαστεί ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 18. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στη συμβασμό 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 28. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Και τώρα να ψηφίσουμε το σύνολο της νομοδότησης. Τελική ψηφοφορία παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Βόν. Εγκρίθηκε η γνωμοδότηση με ευρεία πλειοψηφία. Το επόμενο σημείο είναι οι συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις ε, της ε, συμφωνίας, της συμφωνίας για τις υπηρεσίες της ΤΙΖΑ. Και είχαμε και την γνωμοδότηση πρωτοβουλίας για τις συνεχιζόμενες συγγνώμη, διαπραγματεύσεις στην ΤΙΖΑ, κυρία Βάνα είχε παρουσιάσει την τελευταία φορά 21 Οκτωβρίου ήταν η προθεσμία 65 τροπολογίες έχουν υποβληθεί για την αποτελεσματική απελευθέρωση των του εμπορίου υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες και η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και κυβερνήσεις, Συμβαστικές τροπολογίες έχουν υποβληθεί για τις περισσότερες από αυτές. Η κυρία Βάνα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και θα ε, ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες και τους κοιόδης για την πολύ καλή συνεργασία και την θετική ατμόσφαιρα που είχαμε. Γνωρίζουμε ότι η τίζα είναι αντιφατικό ζήτημα. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί συνένεση υποθέσεων τόσο ριζικά διαφορετικό σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά προσπαθήσαμε πολύ να βρούμε κοινό έδαφος και να έχουμε μια, ένα πνεύμα στην Επιτροπή Ρέτζη σχετικά με τις αρμοδιότητες ε, των τοπικών φορέων και την συνεργασία μαζί τους. Και έτσι είμαστε σε θέση σήμερα να υποβάλουμε ένα κοινό κείμενο. Σας ευχαριστώ. Ας πάμε τώρα στην ψηφοφορία. Ξεκινούμε με την συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 εδώ έχουμε διακριτή ψήφο που ζητάει η συγκήτρια υπέρ στο πρώτο τμήμα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στο δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. We go to amendment 55. Πάμε στην 55. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, 21. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ όχι το συγγνώμη λέει πρόεδρος μου διέφυγε η 48 απερίφθη η 49 και επομένως πρέπει να πάμε 48 ή 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τώρα πάμε στην 50 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική ψήφος άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όχι, όχι, να ελέγξουμε. Την 51 να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική 10 αποσύρεται πρέπει να ψηφίσουμε χωριστά 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα ψηφίζουμε επί της γνωμοδότησης. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Και εγκρίνεται. Ευχαριστούμε κυρία Βάνα. Συγχαρητήρια. Και με αυτό ολοκληρώσαμε με την πρωινή συνάντηση και μπορούμε να προχωρήσουμε με τους συντονιστές αν συμφωνείτε.